Jag är väldigt glad att få hälsa. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να καλωσορίσω θερμά όλους σε, αυτό το απογευμα... σε αυτή την επαγγευματινή πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Να εξηγήσω καταρχήν ότι αν θέλετε να ακούσετε τουρκικά θα παρακολουθήσετε τη διερμηνία από το κανάλι 24 αν θέλετε να παρακολουθείτε την τουρκική γλώσσα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν έχουμε προβλέψει μια δημόσια ακρόαση με γενικό τίτλο «Προοπτική του 2020 για τις γυναίκες στην Τουρκία». Η Τουρκία είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ε, ε, προσχώρησης ε, που ε, συζητείται και λόγω των κριτηρίων της Κοπενχάγης που επίσης συζητούνται σε αυτά τα πλαίσια. Ένα σημαντικό θέμα που ανακύπτει όταν μιλάμε για την προσχώρηση της Τουρκίας είναι η κατάσταση των γυναικών. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή δημόσια ακρόαση επί αυτού ακριβώς του θέματος και θέλω να καλωσορίσω τους ειδικού φιλοξενουμένους μας, τις φιλοξενούμενές μας που ήρθαν για να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να παρουσιάσουν πολύ σοβαρή τεχνογνωσία. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε. Το πρώτο τμήμα των συζητήσεών μας θα αφορά τους στόχους και τις προτεραιότητες για το 2020, στόχοι και προοπτικές για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην Τουρκία στην πορεία προς την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο μέρος της συζήτησης είναι, έχει τον τίτλο «Οι γυναίκες στην Τουρκία ως παράγοντες προόδου. Μέτρα βελτίωσης και βέλτιστες πρακτικές». Αυτές είναι οι γενικές κατηγορίες στα πλαίσια των οποίων θα συζητήσω με τις προοπτικές των γυναικών στην Τουρκία εν ώψη του 2020. Να καλωσορίσω και την εισηγήτριά μας, την κυρία Εμίν Μποσκούρτ. Καλώς ήρθατε. Ξέρω την αφοσίωσή της στο θέμα και την τεχνογνωσία της. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Θα αρχίσουμε και δίνω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στο μέλλον της Τουρκίας και την προοπτική του 2020 εξετάζοντας την κατάσταση στις γυναίκες πώς θα πρέπει να είναι το 2020. Τον περασμένο μήνα ήμουν εισηγήτρια σε μια διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη για την ισότητα των φύλων και είχα την ευκαιρία σε εκείνη τη διάσκεψη να συζητήσω με πολλές γυναίκες από πολλούς τομείς της κοινωνίας της Τουρκίας υπήρχαν και αποκλίνουσες απόψει σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία. Αλλά κάτι στο οποίο συμφώνησαν όλοι είναι ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα για να βελτιώσει την κατάσταση των γυναικών. Γι' αυτό αποφάσισα λοιπόν να δημιουργήσω μια προοπτική του 2020 για τι γυναίκε στην Τουρκία στην έκθεση για να ενθαρρυνώ τι γυναίκε να θέσουν στόχου, οι ίδιε για τον εαυτό του και να δραστηριοποιηθούν συμβάλλοντας προς μια αλλαγή για το καλύτερο. Η Τουρκία σήμερα έχει ένα εθνικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα δράση για την ισότητα των φύλων, αλλά το πρόγραμμα αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική, ούτε θέτει προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων. Αναφέρει μόνο αυτά που ήδη έχουν επιτευχθεί, αντί να προσβλέπει στο μέλλον και τι απομένει να γίνει, ποιες προτεραιότητες πρόκειται να μας απασχολήσουν άμεσα. Έτσι λοιπόν θα συλλέξω απόψεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές από γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους, από ανθρώπους που εργάζονται σε κάθε τομέα επιτόπου. Θα χρησιμοποιήσω τη συμβολή τους για να καταλάβω καλύτερα τα πράγματα, να εντοπίσω προτεραιότητες και να θέσω μέσω και μακροπρόθεσμους στόχους ώστε να έχουμε μια στρατηγική με βιώσιμες συστάσεις ε, για να βελτιώσουμε τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών τώρα και στο μέλλον. Κατά την τελευταία μου επίσκεψη μίλησα με πολλές γυναίκες με επιρροή στη σημερινή αρένα του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και θα σας δώσω ορισμένες απόψεις. Επιφανείς γυναίκες ε, στην Ανατολική Τουρκία που εργάζονται οι πολλές γυναίκες λένε ότι τα βασικά εμπόδια στην απασχόληση είναι πρακτικά στην Τουρκία. Ε, υπάρχουν λίγες εγκαταστάσεις φύλαξης των παιδιών και σύμφωνα με στατιστικές μόνο 1% των παιδιών ηλικίας 0 με 3 ετών βρίσκονται σε κέντρα προσχολικής ε, ε, ηλικίας, οπότε οι μητέρες βρίσκονται στο σπίτι για να τα φροντίζουν και δεν εργάζονται. Πολλές άλλες γυναίκες με ηγετικό ρόλο επιβεβαίωσαν την έλλειψη των γυναικών στη διαδικασία έλλειψη αποφάσεων και το δημόσιο τομέα εν γέννη. Ενώ ο κυβερνητικός τομέας θα μπορούσε να είναι ο πρώτος τομέας που θα έδινε το καλό παράδειγμα για τις, ε, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ισότητας. Αυτά και πολλά άλλα παρουσιάστηκαν ε, σαν ε, γνώμες και συμπεράσματα. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει μακρά ιστορία στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων στην Ευρώπη όταν ε, υιοθέτησε στη δεκαετία του 30 το δικαίωμα ψήφου πολύ πριν από κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι πολλοί νόμοι έχουν ε, θεσπιστεί, όπως ο νόμος για την ισότητα. Ξέρουμε ότι πολλές συμβάσεις και πρωτόκολλα έχουν υπογραφεί, όπως ε, η Σύμβαση ΣΥΝΤΟ για την απάλληψη κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Όμως Γνωρίζουμε επίσης ότι μόνο 9% των εδρών στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση ε, κατέχονται από γυναίκες και 12% αναμένεται να συμβεί στη νέα Εθνοσυνέλευση που θα εκλεγεί τον Ιούνιο περίπου 20% σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις για τα φύλλα, έχει τη θέση 126 η Τουρκία στον κατάλογο μεταξύ 134 χωρών σε ό,τι αφορά το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, ενώ το Ιράν είναι στην 133η θέση πάνω από την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία υπολείπεται και του Ιράν ακόμη εις ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Ξέρουμε επίσης ότι η αναγκαστική ε, γάμη και τα εγκλήματα τιμής ε, είναι πρόβλημα. Οι νεαρές γυναίκες εξαναγκάζονται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο και τελετές ενώ δεν υπάρχει ελάχιστο όριο ηλικίας και δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα που τους παρέχει ο πολιτικός γάμος. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν τεράστιες περιφερειακές διαφορές στην εφαρμογή των νόμων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα στην νομοθεσία, ένα κενό μεταξύ των δικαιωμάτων των παντρεμένων και μη γυναικών και ότι υπάρχει και ένα όριο σε ό,τι αφορά αριθμό ημερών γάμου στις διαζευγμένες γυναίκες. Στην Τουρκία δίνεται μάχη για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, οι γυναίκες που αποτελούν ε, πρότυπα για τη μελλοντική και την ε, τωρινή γενιά και που είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Τώρα, σε σχέση με το μέλλον, στην Ευρώπη υπάρχει η στρατηγική 2020 για την ανανέωση της οικονομίας ε, προτεραιοτήτων που πρέπει να επιτευχθούν πριν από το 2020. Οι υπολογισμοί για την Ευρώπη έχουν γίνει για το 2020 και οι προσδοκίες δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει ε, έλλειψη στο εργατικό δυναμικό. Θα χρειαστεί μέχρι το 2020 όλες τις γυναίκες της η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ω οικονομικό γίγαντα χρειάζεται τι γυναίκε να συμμετέχουν στην απασχόληση και η Τουρκία θα χρειαστεί οι γυναίκε να συμμετέχουν. Η Τουρκία είναι ε, οικονομία σε μεγέθυνση. Το 75% του γυναικείου πληθυσμού όμω δεν συμμετέχει στην, στο επίσημο εργατικό δυναμικό. Συχνά είναι πιο εύκολο οι γυναίκε να κάνουν σταδιοδρομία σε οικογενειακέ επιχειρήσει. Αν όμω μια γυναίκα μπορεί να είναι ενεργητικό, στην οικογενειακή επιχείρηση, γιατί να μην αποτελέσει ενεργητικό και σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. 50% όλων των ε, φοιτητών στα πανεπιστημία είναι γυναίκες. Και τι θα κάνουν αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, θα πάνε να καθίσουν στο σπίτι και να κορνιζώσουν τα διπλώματα και να τα βλέπουν στον τοίχο. Η Τουρκία θα πρέπει να εντάξει, να δραστηριοποιήσει τις γυναίκες, να βοηθήσει τις γυναίκες να βοηθήσουν εκείνες με τη σειρά τους τον εαυτό τους. Αυτό δεν θα ωφελήσει μόνο τις γυναίκες αλλά ολόκληρη την τουρκική κοινωνία. Γι' αυτό αποφάσισα να εργαστώ πάνω σε μια νέα έκθεση για τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, αλλά αυτό με ενοχλεί τώρα που γίνεται. Ίσως μιλούν στην αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να δουλέψω πάνω σε μια νέα έκθεση εξετάζοντας την προοπτική του 2020 για τις γυναίκες στην Τουρκία. Αυτή θα είναι μια προοπτική η οποία οραματίζεται το μέλλον με προοπτική το 2020 και βλέπει ποια θα πρέπει να είναι η ζωή των γυναικών στην Τουρκία που θέτει συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς συνάμα στόχους στέρεα, με, στέρεα μέσα, με benchmark, ορόσημα για να δει ο κόσμος πώς έχει προχωρήσει η Τουρκία στην επιδευσή των στόχων της. Δεν θα το κάνω αυτό μόνη μου. Θέλω να μάθω από τις επιτυχίες των ε, επιτυχημένων γυναικών όπως τις προσκεκλημένες μας να δούμε πώς ε, χειρίστηκαν τα θέματά τους πώς ξεπέρασαν εμπόδια, τι ταμπού έπρεπε να σπάσουν τι έκαναν για να επιτύχουν και θα τις ε, ρωτήσω τι μπορεί να μάθει από εκείνες η τουρκική κοινωνία και θα τους ζητήσω να εντάξουν την εμπειρία του σε μια έκθεση που, θα, που σκοπό έχει να εμπνεύσει άλλε γυναίκε και στην Τουρκία και στην Ευρώπη. Είχα συζητήσει σε πανεπιστήμια με νέε κοπέλε που τώρα αρχίζουν τη σταδιοδρομία του και τι ρώτησα πώ βλέπουν το μέλλον στην Τουρκία, τι προοπτικέ βλέπουν εκείνε για τον εαυτό του στη χώρα αυτή. Ήθελα να του μιλήσω για τα μοντέλα και των ρόλων τους, πώς τα αντιλαμβάνονται. Επίσης ρώτησε τις γυναίκες φίλες μου στο facebook σε σχέση με τους ρόλους ε, ανδρών και γυναικών στην ε, Τουρκία ε, και ανέφεραν διάφορα πρότυπα όπως του, του Πρωθυπουργού και άλλες. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές απόψεις που οδήγησαν σε μια συζήτηση. Οι γυναίκες εξήγησαν τα ε, μοντέλα ρόλο, οι άνδρες πάλι έκαναν ένα διαχωρισμό ε, σε σχέση με πρόσωπα ε, κοσμικά ή μη. Αυτή η πόλωση δημιουργείται από τους άνδρες και έτσι η συζήτηση για την ισότητα των φίλων δυσκολεύεται. Γιατί στο τέλος, σε τελευταία ανάλυση, οι γυναίκες θέλουν να θεωρούνται ίσες. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θεωρούνται ως μέσον Οι γυναίκες στην Τουρκία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον για την καταπολέμηση, ε, για, για, την, για, να, για πολιτικών μαχών που κυριαρχούνται από τους άνδρες. Θα πρέπει να είναι σύμμαχοι στην αλλαγή και οι άνδρες επίσης όλοι να ωφεληθούν από την πρόοδο. Κυρίες και κύριοι γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές δεν ε, γίνονται μια νυχτή, όμως μπορεί να υπάρξει ε, μια διαδικασία πρόοδου. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν τι θα θέλαμε τι θα ευχόμαστε για τις κόρες μας. Αυτό θα πρέπει να ε, ισχύει ε, για αυτό που θέλουμε για όλες τις ε, νέες γυναίκες, σε όλες τις μεγάλες πόλεις και όπου και να ζουν στην Τουρκία. Τους ευχόμαστε ευτυχία, τους ευχόμαστε να γίνουν αυτό που θέλουν. Και για να κλείσω κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ενθουσιώδης σε σχέση με την έκθεση αυτή. Θέλω να δώσω μια νέα προοπτική στις γυναίκες στην Τουρκία. Προσβλέπω στις απόψεις σας, στις εμπειρίες σας και ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ συζήτηση. με ευγνώμων στις ε, συναδέλφους μου εδώ σήμερα και ε, είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία στα πλαίσια του έργου μου για την έκθεση. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Μπόσκοτ για αυτή την εισαγωγή. Έχω τώρα τη χαρά, εξ ονόματος της Επιτροπής μας, να καλωσορίσω την κυρία Λέιλα Κοσκιούν, Γενική Διευθύντρια για την κατάσταση των γυναικών από την Άγκυρα. Κύρια Κοσκούν, ως Γενική Διευθύντρια για την ισότητα των γυναικών ασχολήθηκε με τον συντονισμό και με ευρύτερε ευθύνε για μια σειρά διεθνών δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό, μετέσχευε και στην νομοθετική προπαρασκευαστική δραστηριότητα στην Τουρκία σε ό,τι αφορά νομοθεσίες για, νομοθεσία για θέματα ισότητας. Επιπλέον, μετέσχε σε μια σειρά διεθνών συνεδρίων σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ένωση, αλλά και στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και Υπενθυμίζω απλά στους ε, φιλοξενούμενους μας ότι έχουμε 15 λεπτά maximum χρόνο παρέμβασης για κάθε παρουσίαση. Να επαναλάβω ε, το καλώ ήλθατε και σας δίνω το λόγο αμέσως κύριε Κόσκουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ίσως να μιλήσω λίγο περισσότερο από το τέταρτο. Ζητώ εξ αρχή συγγνώμη. Αγαπητοί σύνδεοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς να εκφράσω τη χαρά μου για την ε, συμμετοχή στη συνάντηση αυτή σήμερα. Με καλέστε να μιλήσουμε για τις προοπτικές ε, εν ώψη του 2020 ό,τι αφορά την ισότητα ανδρών γυναικών στην Τουρκία. Θα σας κάνω λοιπόν μια παρουσίαση για την, ε, το όραμα που έχουμε για την ισότητα εν ώψη του 2020. Θα προσπαθήσω να σας κάνω την παρουσίαση αυτή. Η κυρία Μποσκούτ το υπογράμμισε και αυτή στην ε, εισαγωγή της. Από το 1923 οι γυναίκες στην Τουρκία απέκτησαν δικαιώματα, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά. Η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή, η συμμετοχή τους στην οικονομία ξεκίνησε με την, από την ε, ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ε, βιώσαμε πάρα πολλές ε, κοινωνικές αλλαγές στη χώρα και στην κοινωνία. Από την υποψηφιότητα της Τουρκίας στην Ένωση για ένταξη στην Ένωση και μετά από το 2000 δηλαδή έγιναν πάρα πολλές αλλαγές νομοθετικού χαρακτήρα στο Σύνταγμα και τους απλούς νόμους προστέθηκαν μια σειρά εγγυήσεων νομοθετικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την ισότητα των γυναικών και θα ήθελα να παρουσιάσω τις εξελίξεις αυτές ενώπιόν σας. Δύο φορές άλλαξε το Σύνταγμα, το 2001 και το 2004. Ενισχύσαμε τις εγγύσεις υπέρ των γυναικών, ιδίω το άρθρο 10 αναφέρει ότι οι γυναίκες έχουν είναι ισότιμες με τους άνδρες, έχουν ίσα δικαιώματα, ενώ το δημοψήφισμα που έγινε πέρυσι τον Οκτώβριο του 2010 εισήγαγε στο Σύνταγμα μία νέα πρόταση που λέει, που αναφέρει ότι τι, καμία πράξη δεν μπορεί να αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας. Έτσι βλέπουμε ότι ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των γυναικών. Το 2002 η νομοθεσία τροποποιήθηκε και άλλαξε ο αστικός κώδικας και τροποποιήθηκε η... Βέβαια υπάρχει ακόμα, υπάρχουν ακόμα διακρίσεις σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή, αλλά επί ε, θεωρητικά, δηλαδή στον αστικό κώδικα, δεν υπάρχει καμία διάκριση και σας μπορώ να σας το πω ότι πρόσφατα μετέσχον στις προετοιμασίες της νομοθεσίας για τα δικαιώματα επί των παιδιών, την επιμέλεια. Ε, αυτή τη στιγμή ο νόμος προβλέπει απόλυτη ισότητα. Επιπλέον, η νέα νομοθεσία για την απασχόληση, ένας παλιός νόμος που αναθεωρήθηκε το 2003, προ... απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό το εγγυάται εκ νέου ο νόμος. Επίσης άλλαξε και ο ποινικό κώδικας από το 23, πολλές φορές βέβαια. Τον Ιούνιο του 2005 ο νέος ποινικό κώδικας τέθηκε σε ισχύ και τα εγκλήματα κατά των γυναικών μέχρι τότε εθεωρούνται ως εγκλήματα κατά της κοινωνίας, ενώ μετά το 2005 θεωρούνται ως εγκλήματα κατά ατόμων. Ε, η τιμωρία των, των ε, αδικημάτων αυτών άλλαξε επίσης, επί, ε, αυξήθηκε η ανώτατη ποινή φυλάκισης κατά 50% ενώ ποινικοποιήθηκε και η οικογενειακή βία. Βλέπετε λοιπόν ότι στο επίπεδο του νόμου υπάρχει ισότητα. Η τουρκική νομοθεσία παρέχει μια σειρά εχέγγυων προστασίας της ισότητας. Επιπλέον, η νομοθεσία για την προστασία της οικογένειας που αποσκοπεί στην προστασία της γυναίκας από την συζυγική βία, έννοια που πρωτοεισάχθηκε το 2008 στον νόμο, προβλέπει ότι και τρίτη μπορούν να καταγγείλουν στην αστυνομία ή στις δυνάμεις ασφαλείας περιπτώσεις όπου διαπιστώνουν ότι υπάρχει βία στο εσωτερικό της οικογένειας, ότι ασκείται βία στο εσωτερικό μιας οικογένειας. Σήμερα οι δικαστές επιπλέον έχουν το δικαίωμα να προσανατολίζουν μέλη της οικογένειας σε συγκεκριμένα θεσμικά, σε θεσμικά πλαίσια προστασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα βασικά κείμενα για την ισότητα δικαιωμάτων στην κοινωνία έχει βελτιωθεί. Άλλαξε σημαντικά ε, το νομοθετικό πλαίσιο. Μεταξύ 2007 και 2011 το πέμπτο αναπτυξιακό πλάνο δίνει σημαντική θέση στη γυναίκα για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, της εγγραμματοσύνης τους και υπογραμμίζοντας τις ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό το ένα το προαναπτυξιακό σχέδιο ε, ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Επίσης, στο πρόγραμμα δράσης προβλέπεται να δημιουργηθούν η προστασία καταφύγια για τις γυναίκες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, προβλέπεται να υπάρξει κατάρτιση για το ζήτημα αυτό. Ταυτόχρονα, προβλέπονται δύο προγράμματα δράσης για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και για την ενσωμάτωση των ενιών αυτών στο κέντρο των ε, επερχόμενων νομοθετικών κειμένων. Όπως υπογράμμισε προηγουμένως η κυρία Μποσκούρτ, η Τουρκία ετοίμασε αυτό το πρώτο πρόγραμμα δράση στο ξεκίνημα της δεκαετίας ε, του στο, στο τέλος της δεκαετίας του 90 ε, υλοποιήθηκε αυτό το 98 με συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας. Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα δράσης που ασχολιόταν με το ζήτημα των προβλημάτων των γυναικών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια για τις γυναίκες και στο πλαίσιο πάντα του προγράμματος του Πεκίνου λάβαμε υπόψη και τις διεθνείς συμβάσεις για την την αντιμετώπιση της φτώχειας των ε, γυναικών, την εκπαίδευση των γυναικών, τα μέσα ενημέρωσης. Οκτώ κεφάλαια υπάρχουν για όλα τα θέματα. Συμμετείχαμε στην επεξεργασία όλων αυτών των κειμένων και με την συμμετοχή πολλών ΜΚΟ θέσαμε συγκεκριμένους μέσο και μακροπρόθεσμους στόχους Έχουμε και βραχυπρόθεσμους, πολύ βραχυπρόθεσμους στόχους. Παρακολουθούμε τι γίνεται στο πρόγραμμα δράσης. Κάνουμε δύο ε, συναντήσεις το χρόνο για να βλέπουμε τις εξελίξεις, τις οποίες μετέχουν όλοι οι ε, συνεργαζόμενοι φορείς. Δημοσιεύουμε την έκθεση, τη βγάζουμε και στην ιστοσελίδα μας. Υπογραμμίζουμε τις επιτυχίες. Αύξηση του αριθμού της Σχολική εκπαίδευση των γυναικών, συμμετοχή γυναικών σε δημοτικά σχολεία, κοριτσιών δηλαδή σε δημοτικά σχολεία. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράση. Κάτι άλλο. Η μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Όπως σας είπα, ε, με το 2010 ξεκίνησε μια νέα, ε, ένας νέος προγραμματισμός, τον οποίο μετέχουν όλοι οι κλάδοι της κοινωνίας περιμέναμε να, να υπογράψει η χώρα κάποιες διεθνείς συμβάσεις μεταξύ των οποίων και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τους επόμενους μήνες θα γίνει η υπογραφή. Εγώ εξέτασα την σύμβαση αυτή και βλέπουμε ότι περιλαμβάνει πολλές έννοιες και αρχές που είναι αντίστοιχες με αυτές που ήδη προβλέπει η τουρκική νομοθεσία. Είμαστε απόλυτα αποφασισμένες να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της ε, ενδοοικογενειακής βίας με ενισχυμένο τρόπο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για να επιτευχθεί σε μια κοινωνία δεν αρκεί να υπάρξει αλλαγή νομοθεσία μόνο. Πρόκειται για μια προφανώς απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν νόμοι και εγγυήσεις. Ταυτόχρονα ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτό κάνουμε από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 2000. Χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτό είναι σημαντικό για την Τουρκία και δουλεύουμε και στον τομέα αυτό. Παρά τις πολλές νομοθετικές αλλαγές λοιπόν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες εφαρμογής, χρειάζεται να υπάρξει υποστήριξη από πλευράς κυβέρνησης και χρειάζεται και οι γυναίκες να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιες για τη ζωή τους, να ζητούν να εποφελούνται των δικαιωμάτων τους. Τον τελευταίο καιρό έχουμε προχωρήσει σημαντικά. Οι γυναίκες αυξάν, αυξάνονται τα αιτήματα των γυναικών, γνωρίζουν καλύτερα τον νόμο, τα δικαιώματά τους και έχουν περισσότερες απαιτήσει από τα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της ισότητας. Παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς συμβάσεις και συναντήσεις σχετικά. Ενημερώνουμε τις αρχές στη χώρα μας για τις ε, δραστηριότητες και παρέχουμε πληροφορίες για τις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών στον τομέα αυτό. Ένας σημαντικός τομέας είναι η εκπαίδευση γυναικών και κοριτσιών. Παρά την υφιστάμενη νομοθεσία, βλέπουμε ότι στην Τουρκία τα κορίτσια αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Όταν θέλουμε να δούμε πόσες... Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του αριθμού των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο ανάλογα είναι αγόρια ή κορίτσια. Παρά την, τις διατάξεις του νόμου βλέπουμε ότι ε, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο αριθμός των κοριτσιών που πηγαίνουν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Βλέπουμε επίσης ότι τα, τα μέσα ενημέρωσης και ο ιδιωτικός τομέας έχουν κάνει, ε, ξεκινήσει μια σειρά ε, σχετικών εκστρατιών για να αυξηθεί ο αριθμός των, ε, της ο των γυναικών, των κοριτσιών που πηγαίνουν σχολείο. Σήμερα βλέπουμε ότι ο αριθμός των παιδιών, που, των κοριτσιών που πηγαίνουν σχολείο είναι παρόμοιος με αυτό των αγοριών. Και η πρόοδος αυτή υποστηρίχθηκε πολύ και ενισχύθηκε από τις διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Όπως αυτό που λέμε, κορίτσια πάμε σχολείο. Άλλα παραδείγματα. Έχουμε πολλούς, πολλοθεσμικά όργανα που με το ζήτημα της ισότητας. Και θέσαμε ένα στόχο αύξησης της εγγραμματοσύνης των γυναικών άνω των 15. Εκατοντάδες γυναίκες μάθανε να διαβάζουν και να γράφουν χάρη σε αυτή την ειδική εκστρατεία. Μετά, το σχετικό πλαίσιο πρόγραμμα του προγράμματος του ΟΗΕ για την ανάπτυξη. Υπάρχει πρόγραμμα για, ειδικό πρόγραμμα για αύξηση του ποσοστού ε, ε, ε και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυξήσεων ξεπερνάει άλλες χώρες όπως το Μπαχρέιν και φτάνει σε επίπεδα Γερμανίας. Επίσης, θέλουμε να αφαιρέσουμε από τα σχολικά εγχειρίδια όλα τα, ε, όλες τις εξιστικές ε, νοοτροπίες. Προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε τα σχολικά εγχειρίδια βγάζοντας κάθε φράση που μπορεί να οδηγήσει σε διακριτική αντιμετώπιση και που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα βιβλία. Μια άλλη σημαντική διάσταση στο θέμα ισότητας αφορά την απασχόληση, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία και τη μείωση της γυναικείας φτώχειας. Στο πλαίσιο της, εναμέ, της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, ε, υιοθετήσαμε μια σειρά κειμένων για την αξιολόγηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση. Ε, μεταξύ των προτεραιοτήτων υποστηρίζουμε γυναίκες που θέλουν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση και δουλέψαν πολύ στον τομέα αυτό. Βάσει στοιχείων του 2009, στην Τουρκία η συμμετοχή των γυναικών στην, ε, ναι, στην ε, ενεργή οικονομική δραστηριότητα είναι 22%. 26% των γυναικών που είναι σε ηλικία εργασίας δουλεύουν. Υπάρχει μία ε, ε, έξοδος από την Ήπεθρο. Οι γυναίκες στην Τουρκία, που σημαίνει ότι οι γυναίκες ε, των χωριών δεν αισθάνονται ε, σε θέση να δουλέψουν στις μεγάλες πόλεις, μένουν αποκλεισμένες, μένουν έξω από τον επίσημο κόσμο της εργασίας ή δουλεύουν σε ανεπίσημα, παράλληλα, σε ανεπίσημες και παράλληλες δομές. Χρειάζονται και άλλα μέτρα για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν μια σειρά προγραμμάτων για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας οργανισμός πρόφησης της γυναικής απασχόλησης που προχωρεί σε επαγγελματική κατάρτιση γυναικών. Βλέπουμε ότι όσες μετέχουν σε τέτοια μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, μάλλον από όλες αυτές, 40 με 60% επιτυγχάνουν. Παίρνουν πτυχίο και έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη βάσει μιας τελευταίας νομοθεσίας. Τον Φεβρουάριο του 2011 υιοθετήθηκε ένας νέος νόμος σχετικά, ενώ ένας άλλος νόμος του 7 προβλέπει ότι ορισμένα προϊόντα που θεωρούνται προϊόντα που παράγουν οι γυναίκες που μετέχουν, στα, που μετέχουν στα προγράμματα αυτά μπορούν να πολιθούν χωρίς ΦΠΑ αφορολόγητα και οι γυναίκες που βρίσκουν ε, μισθωτή εργασία με πέντε χρόνια μετά το τέλος ε, της εκπαίδευσης αυτής μπορεί να πληρωθούν, να μειθούν χωρίς φορολόγηση του μισθού τους. Όλα αυτά για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην ε, αγορά εργασία. Επίση υπάρχουν και νέε ε, διατάξει για την. Ε, ε τις να προχωρήσω πιο γρήγορα γιατί έχω πολλά ζητήματα. Στο θέμα της εκπαίδευσης υπάρχουν και μια σειρά ιδρυμάτων που παρέχουν ενίσχυση και συμβουλευτική για τις γυναίκες που να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ειδική υποδομή για τις γυναίκες που ασχολούνται με αγροτικές δραστηριότητες. Πολιτικός τομέας τώρα, το ανέφερε η κυρία Μποσκούρτ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη, περισσότερα αιτήματα συμμετοχή στην πολιτική ζωή από πλευράς γυναικών. Στι στις του 2011 θα υπάρχουν πιστεύουμε περισσότερες, πολύ περισσότερες γυναίκες βουλευτές. Κάτι άλλο. Βία κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό αδίκημα. Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά δραστηριοτήτων σχετικά. Δυστυχώς δεν λάβαμε. Δεν είχαμε ακόμα σημαντική επιτυχία. 15% των γυναικών αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο στην Ήπεθρο. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, σας είπα ότι πέρασαν πολλοί νόμοι που προσπαθούσαν να καταπολεμήσουν την συζυγική βία, αλλά στην εφαρμογή του νόμου πάσχει. Είμαστε όμως αποφασισμένες να αγωνιστούμε κατά της μάστιγας αυτής. Πρέπει να αλλάξει ακόμα κάπου η νομοθεσία. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των ε, ιερωμένων για να μπορούν να κατευθύνουν ευκολότερα και καλύτερα τις γυναίκες στα καταφύγια που είναι, ε, όταν είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ξέρουμε τα προβλήματα των γυναικών στην Τουρκία, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και το κράτος συνολικά, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, όλοι οι τομεί της κοινωνίας δουλεύουν με έντονο τρόπο για να μπορέσουν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα των γυναικών και είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τις γυναίκες. Είμαστε δε πεπισμένοι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας υποστηρίξει στι προσπάθειές μας. Ευχαριστώ εκ νέου για την ε, υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Τσόσκουν. Εξ ονόματος τώρα της ευρωπαϊκή Επιτροπής θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Στέφανο Σανίνο, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής από την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη συνεδρία σε αυτή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τις παρατηρήσεις της γυναικής διευθύντριας για τον ρόλο των γυναικών και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Τουρκία όσον αφορά τον ρόλο που διδραματίζουν οι γυναίκες. Θα ήθελα λοιπόν εξ αρχής να πω ότι ήδη από το 1998 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να υποβάλλει συστηματικά εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο που είχε σημειωθεί στην Τουρκία για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των γυναικών και της τουρκικής κοινωνίας, έκτοτε λοιπόν έχουμε καταφέρει να δούμε ένα σημαντικό αριθμό σημαντικών πρόοδων που έχουν επιτευχθεί. Θα έλεγα ότι η πρόοδος αυτή είναι ενδεχομένως κάπως αργή, αλλά τουλάχιστον σταθερή και όπως είπε η Γενική Διευθύντρια έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα στον τομέα της εφαρμογής το σημαντικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε ότι το ζήτημα των φύλων στην Τουρκία παραμένει ένα ζήτημα πρόκληση από πάρα πολλές πτυχές. Υπάρχουν δύο στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία τονίστηκαν. Το ένα έχει να κάνει με την εκπαίδευση και το δεύτερο έχει να κάνει με την αγορά εργασίας. Ο πόντος αληθεύει ότι δυστυχώς η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι μία από τις χαμηλότερες στις χώρες του ΟΣΑ και οι γυναίκες επηρεάζονται ιδιαίτερα από το υψηλό ποσοστό μη καταχωρημένης, μη δηλωμένης εργασίας, ιδίως στον γεωργικό τομέα, στις αγροτικές περιοχές, στην Ήπεθρο, όπου πολλές φορές εργάζονται στα πλέγια οικογενειακών επιχειρήσεων και όπου πολλές φορές η αδήλωτη αυτή εργασία φτάνει το 40%. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ζήτημα στο οποίο δεν είχαμε πολύ θετικέ εξελίξεις. Το χάσμα ανάμεσα στα φύλλα τα δύο φύλλα όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει πια μειωθεί, θα λέγαμε ότι έχει κλείσει εντελώς, αλλά όσον αφορά τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα, μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία νομοθετικά κάποια νομοθετήματα, σχέδια δράσεις τα οποία έχουν ε, υιοθετηθεί από την κυβέρνηση και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Καταρχάς, το σχέδιο δράσης για την ισότητα των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών για την περίοδο 2008-2013. Σχέδιο δράσης το οποίο μας αφορά γιατί όντως υπογραμμίζει τα προβλήματα συμμετοχής ε, των γυναικών καθώς επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι γυναίκες στην κοινωνία Δυστυχώς, οι ανθρώπινοι και χρηματικοί πόροι που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο δράσης δεν αρκούν. Επίσης πιστεύουμε ότι ε, όσον αφορά τους μετρήσιμους στόχους, ακόμα το σχέδιο αυτό δεν είναι απόλυτα σαφές. Επίσης είχαμε μία εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, η οποία διενεμήθηκε έχει ως στόχο την πρόθεση της απασχόλησης των γυναικών και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του στην αγορά εργασίας. Και υπάρχει και ένα Εθνικό Συμβούλιο για το συντονισμό των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την απασχόληση των γυναικών. Πιστεύουμε ότι αυτό το μέσο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Τουρκία. Το ίδιο ισχύει και για την θέσπιση μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες στο τουρκικό κοινοβούλιο επιτροπή η οποία είναι σημαντική και θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα νομοθετήματα εκείνα, την νομοθετική εργασία που πρέπει να γίνει προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η εθνική νομοθεσία με τις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης πιστεύουμε ότι ε, το τριμερές πρωτόκολλο το οποίο έχει συναυθεί ανάμεσα στις κοινωνικές υπηρεσίες, την Υπηρεσία Προστασίας των Παιδιών και τη Γενική Διεύθυνση για την Κατάσταση των Γυναικών με την ε, υποστήριξη της, ε, των τουρκικών αστυνομικών δυνάμεων είναι κάτι το πολύ σημαντικό γιατί θα βοηθήσει τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τις γυναίκες και τα παιδιά που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Μέσω αυτών λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν ε, ήδη κάποια νομοθετικά στοιχεία τα οποία έχουν εγκριθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα. Αυτό που θα ήταν όμως ιδιαίτερα χρήσιμο ήταν, ε, θα ήταν να δούμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών με μια μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, ενώσεων, των συλλόγων γυναικών. Ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον τομέα αυτό υφίστανται ακόμα σημαντικά προβλήματα και σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το ότι ε, η νομοθεσία όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένε διατάξεις που θα μπορούσαν ε, να οδηγήσουν σε μια πιο επαρκή πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών στην τουρκική πολιτική ζωή και γενικότερα στην τουρκική δημόσια ζωή και η συμμετοχή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή και οι υψηλόβαθμες θέσεις στην δημόσια διοίκηση δεν προορίζονται τόσο για τις γυναίκες. Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Προβλήματα επίσης εντοπίζονται στα εγκλήματα τιμής, στην ενδεκογενειακή βία, καθώς επίσης και στους αναγκαστικούς γάμους. Έχουμε κάποια στατιστικά δεδομένα τα οποία δυστυχώς, δυστυχώς καταδεικνύουν την ε, σοβαρότητα του φαινομένου αυτού. 39% των ε, γυναικών δηλώνουν ε, ότι ήταν θύματα συζυγικής βίας και ένα 13% ήταν θύματα σεξουαλικής βίας. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ακόμα τα, δεν προβλέπονται, προβλέπεται το απαραίτητο πλαίσιο στη χώρα προκειμένου οι γυναίκες να μπορούν εύκολα να καταφεύγουν στην αστυνομία ή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες περιπτώσεις αυτές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους και θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες στους τομείς αυτούς. Όσον αφορά την ε, ενδοοικογενειακή βία, έχουν αρχίσει να επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια ήδη πολύ σημαντικές κυρώσεις, ιδίως όσον αφορά τα εγκλήματα τιμής και τις δολοφονίες τιμής. Πιστεύουμε πάντως ωστόσο ότι θα πρέπει η πρακτική αυτή να γίνει ακόμα πιο διαδεδομένη, γιατί ε, η όλη διαδικασία προσφυγής στο δικαστήριο και επιβολής κυρώσεων δεν εφαρμόζεται ακόμα με τρόπο ιδιαίτερα σταθερό. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το ζήτημα της ε, κατάρτισης των ε, αρχών επιβολής του νόμου, καθώς επίσης και των ε, δημοσίων θεσμικών αρχών, οι οποίες στάσονται κατά της ε, βίας κατά των γυναικών. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυξάνονται επίσης τα εγκλήματα και δολοφονίες τιμής και τα καταφύγια για τις γυναίκες, καθώς επίσης και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας των γυναικών ακόμα περιορισμένες. Επίσης, αναφερθήκατε στο ζήτημα των σχολικών εχειριδίων τα οποία αυτή τη στιγμή θέλετε να προσαρμόσετε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε κάποια στερεότυπα τα οποία υφίστανται ακόμα σε ορισμένα σχολεία. η διαδικασία ένταξης, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό μέσο επίτευξης πρόοδου όσον αφορά το ζήτημα της ισότητας των φύλων στην Τουρκία. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα κεφάλαια στο κοινοτικό κεκτημένο, τα οποία έχουν να κάνουν με το ζήτημα των φύλων, το κεφάλαιο που έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση και που καλύπτει και τα ζητήματα καταπολέμησης των διακρίσεων ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και έχουμε και ένα κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά συγκεκριμένε δράσει για τον τομέα αυτό. Ε, έχουμε έπειτα το κεφάλαιο 23 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαστικό σύστημα, το οποίο επικεντρώνεται στην ισότητα των γυναικών, τα δικαιώματα των γυναικών, ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, καταπολέμηση της ενδεκογυναικής βίας, πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών και έχουμε συγκεκριμένα δύο διεθνή νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με την ενδοκογενειακή βία, την δήλωση των Ηνωμένων Εθνών κατά της βίας κατά των γυναικών, καθώς επίσης και το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Και υπάρχει και ένα τρίτο κεφάλαιο, το υπαριθμό 24, για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, το οποίο ασχολείται πιο συγκεκριμένα με την εμπορία ανθρώπων και περιλαμβάνει κάποιες διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα αυτό συμπεραβαλλομένης της σύμβασης και της δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ε, ανθρώπων. Δυστυχώς αληθεύει ότι ε, χθες είχαμε την 401η ε, συνάντηση του Συμβουλίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, του Συμβουλίου Σύνδεσης και είπαμε ότι καθυστερούν οι διαπραγματεύσεις Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στην πολιτική βούληση που εκφράζουν και οι δύο πλευρές και δυστυχώς αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε γρήγορα στην ενταξιακή διαδικασία. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του επηρεάζει το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Κάποιες θετικές τώρα εξελίξεις ε, στη σχέση με την Τουρκία. Έχουμε σημαντική χρησιμοποίηση χρηματοδοτικής βοήθειας που, ε, παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο. Και έχουμε και κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, θα ήθελα να φερθώ σε κάποια από αυτά, τα οποία έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν και να προκαλέσουν κάποιες σημαντικές νομοθετικές τροποποίησεις που αν εφαρμοστούν πλήρως και το ζήτημα της εφαρμογής της υλοποίησης είναι κάτι πολύ σημαντικό όπως είπατε και εσείς, θα μπορούσαν να επηρεάσουν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, συμβάλει πολύ στην χρηματοδότηση και τη διαμόρφωση δύο εθνικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και για την πρόθεση της ισότητας των φύλων. Επίσης ε, έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό προγραμμάτων που υπάγονται σε αυτό το σχέδιο δράσης και τα οποία έχουν ε, εγκριθεί από κοινού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Θα ήθελα απλώ να αναφερθώ σε κάποια από τα προγράμματα αυτά, μόνο και μόνο για να σας δείξω ποια είναι το είδος συνεργασίας που έχουμε. Έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα για την πρόθεση της ισότητας των φύλων, πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να ενδυναμωθούν οι ικανότητες της Γενικής Διεύθυνσης για την κατάσταση των γυναικών, καθώς επίσης και όλων των άλλων παραγόντων εκείνων που βοηθούν την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της γενικότερης μάχης της γενικότερης καταπολέμησης της ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για τη δημιουργία καταφυγίων για τις γυναίκες εκείνες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Οχτώ πλήρη τέτοια καταφύγια έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας. και προσπαθήσαμε επίσης να ευαισθητοποιήσουμε και τις γυναίκες για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης εργαζόμαστε ιδιαίτερα έντονα για την ενδυνάμωση, χειραφέτηση των γυναικών, για την ενδυνάμωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων υπέρ των γυναικών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Τουρκίας και θέλουμε να έχουμε μία προσέγγιση ευαίσθητοι ως προς τα φύλλα σε στις κοινωνικές εκείνες υπηρεσίες που παρέχονται από, όλους, από όλες τις βαθμίδες της διοίκησης σε τοπικό επίπεδο καθώς επίσης και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε το ζήτημα της απασχόλησης των γυναικών. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες υπέρ των γυναικών σε τοπικό επίπεδο ιδίως όπου νομίζω ότι ιδίω στις λιγότερο αναπτυγμένες ε, περιοχές της ε, χώρας είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις γυναίκες να καταφέρουν να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες ε, θέσεις εργασίας και να ξεπεράσουν τα προβλήματα εκείνα, τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης θέλουμε να αυξήσουμε την καταχώρηση, την εγγραφή των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος εδώ είναι να ευνοήσουμε τις εγγραφές, να μειωθεί ο αριθμός των κοριτσιών που εγκαταλείπουν το σχολείο, να δώσουμε στις γυναίκες, στα κορίτσια καλύτερες, καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου στη συνέχεια να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και θέλουμε να αυξήσουμε επίσης και τη συνειδητοποίηση των ίδιων των γονιών για το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση για τα κορίτσια. Τέλος, όσον αφορά την εκπαίδευση πάλι, να σας πω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά την πρόθεση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Όλα αυτά αποτελούν τμήμα απλώς της εργασίας που κάνουμε από κοινού με τις τουρκικές αρχές τα αριθμητικά στοιχεία είναι κάπως ε, άψυχα θα έλεγα, ψυχρά, αλλά είναι σημαντικά προκειμένου να καταφέρουμε να σας καταδείξουμε τι ακριβώς κάνουμε. 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δίνονται στα προγράμματα αυτά, ένα πολύ σημαντικό ποσό για τον συγκεκριμένο αυτό τομέα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, η κοινή μας αυτή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική προκειμένου να καταφέρουμε να τονώσουμε και την ίδια την Τουρκία, προκειμένου να κινητοποιηθεί και η Τουρκία να εγκρίνει την καθολική αυτή αρχή της ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, πιέζουμε για την ε, μεταφορά και την εφαρμογή, την υλοποίηση της ε, νέας κοινωτικής νομοθεσίας στον τομέα αυτό, που αποτελεί για μας ε, σημαντική προτεραιότητα και θέλουμε να μέσω της κοινωτικής χρηματοδότησης να βοηθήσουμε την Τουρκία στις προσπάθειες της αυτές. Να τονίσω επίσης ότι η επιβολή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων αποτελεί πολύ σημαντική προϋπόθεση για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως σας είπα ήδη από το 1999 παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις όλες τις εξελίξεις και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες που είχε καταβάλει η τουρκική κυβέρνηση και η τα άλλα θεσμικά όργανα, καθώ επίση και η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, προκειμένου να δοθεί ένα υψηλότερο επίπεδο βιωσιμότητας στο γενικότερο αυτό σχέδιο της χειραφέτησης και της ενδυνάμωσης των γυναικών, παρέχοντάς τους καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη κατάρτιση, καλύτερες θέσεις εργασίας και απαλλάσσοντάς τις από την ενδοκογενειακή βία και την εμπορία. Σας ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σανίνο για την ε, συνεκτικότατη αυτή παρουσίαση της ε, παρακολούθησης των κριτηρίων της Κοπενχάγης που άρχισε το 1988. Πολλά προβλήματα επίσης από ό,τι φαίνεται ανέκυψαν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που θεσπίστηκε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής που παρευρίσκονται και συνεργάζονται με την εισηγήτρια Πέντε λεπτά χρόνο ομιλίας έχει κάθε βουλευτής σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Η κυρία Μποσκούρτ, η συγγήτρια, έχει πρώτη το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή, γι' αυτό έχω και πολλές ερωτήσεις. Άκουσα πολλά στοιχεία, εγώ ανέφερα το 2020 ως ημερομηνία, ακούσαμε και άλλες. Μιλήσαμε, εσείς μιλήσατε για το 2023 που και αυτό είναι το σημαντικό γιατί είναι τα 100 χρόνια της ύπαρξης της τουρκικής δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι βάζετε αυτή την ε, ημερομηνία σαν ορόσημο σε σχέση, τι, τι όραμα είναι αυτό που έχετε συγκεκριμένα για το 2023 σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης η βία, είναι τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία η βία κατά των γυναικών. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν ότι τρεις γυναίκες την ημέρα χάνουν τη ζωή τους ε, ως θύματα βίας. Τι μπορεί να γίνει εδώ συγκεκριμένα. Ακούσαμε για πολλέ, πολλούς νόμους που ε, υπάρχουν, αλλά στην πράξη πώς εφαρμόζονται. Επίσης, ε, εδώ και χρόνια υπήρξε η εγκύκλειος για την καταπολέμηση της βίας. Αναφέρθηκε και ένα ταμείο για τις γυναίκες, ώστε να υπάρχουν τα διαθέσιμα οικονομικά κονδύλια για όλες αυτές τις δράσεις. Ε, υπάρχει αυτό το ταμείο, πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα, τι κάνει ή αν δεν λειτουργεί, γιατί όχι. Επίσης, ε, μία ερώτηση για τα ψηφοδέλτια. Ε, οι εκλογές 12 Ιουνίου. Ε, υπάρχουν πολλές γυναίκες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια γιατί βγήκαν. Αν δούμε όμως τις εκλογικές περιφέρειες, οι πιθανότητες εκλογής των γυναικών είναι περίπου 12%. Δεν είναι μεγάλες οι πρόοδοι. Από 9 πήγαμε στο 12%. Ίσως ο στόχος δεν είναι αρκετά φιλόδοξος. Τι ακριβώς γίνεται για να αλλάξουν τα πράγματα. Υπήρξε ένα δημοψήφισμα για τη θετική διάκριση και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι υπέρ των μέτρων διακριτικής μεταχείρισης θετικής υπέρ των γυναικών. Τι γίνεται για να περάσουν στην πολιτική περισσότερες γυναίκες. Σε κάθε έκθεση συζητούμε τα ίδια προβλήματα είναι κάτι που τα ακούμε ξανά και ξανά. Αλλά μέχρι τώρα σκοντάφτει το πράγμα. Δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα ούτως ώστε να περάσουν σε θέσεις ε, υπεύθυνε οι γυναίκες στη λήψη των αποφάσεων. Όταν μιλάμε για ένα όραμα, για μια στρατηγική, τι ε, βασικές προτεραιότητες θα αποφασίσουμε για τη στρατηγική αυτή. Ποιες είναι οι βασικές δράσεις για να δουλεύουν περισσότερες γυναίκες. Είναι μικρό το ποσοστό ακόμα στην αγορά εργασίας και τι πρέπει να γίνει για να πετύχουμε τους στόχους μας μέχρι το 2020 ή το 2023. Ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ. Η επόμενη ομιλήτρια η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους τις εμπειρογνώμονες για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Συγγνώμη που άργησα και έχασα το πρώτο κομμάτι. Ελπίζω πραγματικά η προοπτική του 2020 για τις γυναίκες στην Τουρκία να είναι μια ευρωπαϊκή προοπτική. Εγώ είμαι θερμή υπέρμαχος της ένταξης της Τουρκίας στην Ένωση εφόσον θα έχει υιοθετήσει ε, όλο το κυριακτημένο η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία νομίζω ότι θα ωφεληθούν πάρα πολύ από τη διαδικασία αυτή αλλά και από την ίδια την ένταξη. Βέβαια, στα πλαίσια του 2020 έχουμε υπόψη μας και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και εμείς για τη δικιά μας προοπτική του 2020 τις Γυναίκε της Τουρκίας γιατί έχουμε γυράσκοντα πληθυσμό και πολλές κενέ θέσεις που πρέπει να πληρωθούν τα επόμενα 10-15 χρόνια και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έρθετε στη Δύση να καλύψετε κάποιες κενές θέσεις εσείς από την Τουρκία και σε οικονομικό επίπεδο είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί εσείς οι γυναίκες είστε αγοραστικό κοινό, πολυπληθές κοινό και θα ήταν αμοιβαία εποφελές κάτι τέτοιο. Δυστυχώς υπάρχει όλο και περισσότερο σκεπτικισμός, άνθρωποι που αντιδρούν στην ιδέα της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας. Και θέλουν να επιμένουν σε αυτά που ακόμη δεν βαίνουν καλό στην Τουρκία και συχνά τα δικαιώματα των γυναικών χρησιμεύουν ε, ως παράδειγμα και επιχείρημα για να ισχυριστούν η, ισχυριστεί η μερίδα αυτή ότι η Τουρκία δεν πρέπει να προσχωρήσει. Γι' αυτό όμως εγώ είμαι υπέρ της διαδικασίας προσχώρησης, γιατί αυτό θα είναι καταλήτης αλλαγής. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τις ε, εμπειρογνώμονες από την Τουρκία. Σε ποιο βαθμό είναι αλήθεια και κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο ρόλος της ε, ένταξης για αλλαγές υπέρ της χειραφέτησης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή προοπτική θα συνέβαιναν όλα αυτά, οι βελτιώσεις. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει η ευρωπαϊκή προοπτική για σας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κορνέλισεν. Και τώρα η κυρία Γιανακουδάκη παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία, κυρίες μου. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας πείτε τις σκέψη σας. Καταρχήν να συγχαρώ την νησηγήτρια, η Μεσκιώδης. Η προσέγγιση της είναι εξαιρετική, καλύπτει ευρύτα τους τομείς με πολύ ενδιαφέροντα και ωραίο τρόπο. Και το Facebook καλό μέσον είναι, αλλά όσε δεν έχουν Facebook, αυτές είναι που θέλουμε να φτάσουμε. Και βεβαίως οι γυναίκες των ομάδων των μειονοτήτων. Αργότερα θα τα δούμε και αυτά. Οι ομιλητέ είπαν ότι βελτιώθηκαν πολλά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία και πριν από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ε, ε, ε, πριν από τη Θάτσερ είχαν ε, προηγηθεί υπάρχουν τομείς βελτίωσης δεν θα επισέλθω σε όλους τους σχετικούς τομείς αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Τουρκία είναι κυρίαρχο κράτος με πολιτιστικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές που πρέπει να τις σεβαστούμε και να δουλέψουμε στα πλαίσια τους προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. Θα πρέπει να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στις διαφορετικές περιοχές γιατί η Άγκυρα έχει πιο μορφωμένες γυναίκες από ό,τι είναι οι γυναίκες στην Ήπεθρο. Ως ε, Βρετανίδα Ευρωβουλευτής ε, προσεγγίστηκα σε τρεις τομείς από γυναίκες από την Τουρκία. Καταρχήν, ε, τις γυναίκες από την Τουρκία και την περιοχή των Κούρδων. Επίσης έχουμε στο Λονδίνο την Ένωση των Γυναικών Ρότσα που επίσης είναι ένας σύλλογος ε, γυναικών από την Τουρκία που ήρθαν να συζητήσουν μαζί μου το θέμα της βίας που αντιμετώπισαν οι πολιτικές ακτιβίστριες από τις δυνάμεις ασφαλείας, πιστεύω, της Τουρκίας, συμπεριλαμβάνοντας ε, και περιπτώσεις βιασμών πολλές. Και μια άλλη ομάδα δεν είναι τεχ... τουρκική κανονική αλλά τουρκοκυπριακή ομάδα, δηλαδή γυναίκες που ζουν στα, στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα ενός κράτους μέλους της Ένωσης. Μην ξεχνάμε τις τουρκοκύπριες γυναίκες που θέλουν την ελευθερία τους το ταχύτερο δυνατόν. Χαιρετίζουμε λοιπόν την παρουσία σας εδώ και Θέλουμε να ενταχθεί στην Ένωση Τουρκία το ταχύτερο δυνατόν. Ό,τι ακούσαμε είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αλλά υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης. Και νομίζω ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Και ελπίζω κατά την πορεία αυτή να σας στηρίξουμε και να στηρίξουμε τις γυναίκες. Εσείς τι θα κάνετε για τις ομάδες των μειονοτήτων που προανέφερα. Πόσο ασφαλείς και προστατευμένες είναι οι γυναίκες όταν εισάγεται αλλαγέ, ε, αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά σε τελευταία ανάλυση εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε ασφαλείς και εσείς στην Άγκυρα είστε ασφαλείς και όλοι είμαστε ασφαλείς στα σπίτια μας, αλλά στα χωριά ε, όταν κλείνει η πόρτα και είναι αντιμέτωπη η γυναίκα με τον άντρα, ο άντρας μπορεί να είναι δυσαρεστημένος με όλα αυτά. Μπορούμε να τις υποστηρίξουμε και τις γυναίκες. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες που δεν είναι τόσο κοντά στις δικές μας ασφαλείς περιοχές. Και πάμε έτσι στην Ήπεθρο, όπου θα πρέπει να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι η τρεις τομείς που ήθελα να καλύψω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιανακουδάκη. ξεκίνησε η συζήτηση τώρα. Όσοι συνάδελφοι, όσοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν, παρακαλώ μεταξύ των, των ομιλητριών πρώτα κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές γιατί τη πολύ ενδιαφέρουσα και εκτεταμένη παρουσίαση των εξελίξεων στην Τουρκία και νομικά αλλά και ουσιαστικά και τι κάνει η Επιτροπή σας. Δύο θέματα θέλω να αναφέρω. Ο κύριος ε, Σανίνο μίλησε για το μικρό ρυθμό γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό κατά την άποψή μου είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, η ενδοοικογενειακή βία και οι άλλε μορφέ βία κατά των γυναικών βρίσκονται σε ψηλό επίπεδο. Το ότι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες οι γυναίκες και άρα δεν μπορούν να ζήσουν τη δική τους ζωή αλλά εξαρτώνται από τον σύζυγο, τον πατέρα, τον συγγενή τέλο πάντων που τους ε, κρατάει στο σπίτι υπό την βία. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτών. Επίσης ως Ένωση πρέπει να, έχουμε, ε, να υποστηρίξουμε τις οργανώσεις των γυναικών που αγωνίζονται κατά της ενδοοικογενειακής βίας ή των αγκαστικών γάμων, αλλά και η οικονομική διάσταση είναι μια, η οικονομική ελευθερία είναι μια άλλη διάσταση. Επίσης, το θέμα του επίπεδου εκπαίδευσης, αυτό αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των γυναικών που μετέχουν στην εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο παρέμεινε ίδιος, αυξήθηκε, μειώθηκε. Υπάρχει μια σχέση μια γυναίκα για να είναι εξάρτητη και να βρει δουλειά και να είναι εξάρτητη και συναισθηματικά σχετίζεται και με την παιδεία. Κάτι άλλο που ανέφερε η κυρία συνάδελφος. Τις πολιτιστικές και θρησκευτικέ διαφορές που πρέπει να σεβαστούμε. Εγώ πάντα έχω επιφυλάξεις όταν μιλάμε ιδίω για θέματα δικαιώματα της γυναίκα, δικαιωμάτων της γυναίκας. Βεβαίως πρέπει να σεβόμαστε τις παραδόσεις. Και η Τουρκία επίσης το δέχεται δέχεται το οικουμενικό δικαίωμα της του αυθύπαρκτου δικαιώματος δικαιώματος ε, και της ελευθερίας των γυναικών, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικέ ελευθερίες. Και αυτό θέλουν να υποστηρίξουμε εμείς και οι γυναίκες στην Τουρκία. Από τη δική σας πλευρά, τι κάνετε. Πώς αντιμετωπίζετε περιπτώσεις που υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ αυτών που κάποιοι αποκαλούν πολιτιστικά και θρησκευτικά αιτήματα και της, του ευρύτερου πλαισίου των δικαιωμάτων της γυναίκας που είναι μια μόνιμη αιστεία αμφισβήτησης και σε εμά. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Η κυρία Μπάουερ. Πολλές πληροφορίες είχαμε. Λέμε πολλές φορές ότι στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλος δρόμος μεταξύ της νόμο και έργο ισότητας. Η απόσταση αυτή φοβάμαι στην Τουρκία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα που δεν τέθηκαν προς το παρόν. Αν θυμάμαι καλά, από μία επίσκεψή μας στην Τουρκία πριν λίγα χρόνια, είδαμε κάποιες, κάποια συνήθιστα προβλήματα για για την καταχώρηση των ληξιακών πράξεων γεννήσεως των, των κοριτσιών που έχει συνέπειες και στην ε, εγγραφή στα δημοτικά των κοριτσιών. Μετά την ε, επίσκεψή μας, από ό,τι κατάλαβα, ξεκίνησε μια καμπάνια και υπήρξαν πληροφορίες ότι 20.000 κορίτσια καταχωρήθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα. άλλαξε η κατάσταση, υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφορές μεταξύ των καταχωρήσεων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των κοριτσιών στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τουρκίας. Η, τα εγκλήματα τιμής τώρα είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Η κατάσταση τώρα σε αυτό το τομέα ιδίω μεταξύ της νομικής πραγματικότητας και της ουσιαστικής πραγματικότητας είναι τεράστια. Γιατί για πολύ μεγάλο διάστημα ο ποινικό κώδικας περιελάμβανε την ως έγκλημα αυτό το, τα εγκλήματα τιμή. Παρά τα αυτά η υλοποίηση της νομοθεσίας ε, είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη. Τι προτίθεστε να κάνετε, τι σχεδιάζετε να κάνετε για το ζήτημα αυτό στη στρατηγική σας. Τρίτη ερώτηση. Όταν πήγαμε στην Τουρκία κατάλαβα ότι η ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα γυναικών στέκονται σε αδύναμες βάσεις. Υπήρξαν αλλαγές. Τελευταία ερώτηση. Αν κατάλαβα, κατάλαβα καλά, τις επόμενες μέρες ξεκινά μια, ένα συνέδριο, μια διεθνής διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη για τα δικαιώματα για τις, κατά της ε, θα συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή με μια καμπάνια αύξηση της επίγνωσης ε, ευρύτερα για την καταπολέμηση της βίας. Eh, Ευχαριστώ. Η κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω ασχοληθεί 9 χρόνια με το θέμα των εγκλημάτων τιμής. Ήμουν και στο Συμβούλιο της Ευρώπης στην ίδια ομάδα και παρακολούθησε και την ε, τουρκική συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την εμπορία. Θέλει πολύ καιρό η Τουρκία για να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα γιατί βλέπουμε ότι τα εγκλήματα τιμής δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζονται. Προσωπικά Πήγα πρόσφατα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και την Αντιόχεια. Και είδα τεράστιες διαφορές στα επίπεδα ζωής και στην οτροπία του κόσμου. Είδα τεράστιο αριθμό αγράμματων γυναικών ή κούρδων γυναικών. Κάτι εξαιρετικά προβληματικό. Είναι πολύ δύσκολο να τηρήσει η Τουρκία τους ευρωπαϊκούς στόχους της ε, και την στρατηγική της Ευρώπης εν ώψη του 2020 με τόσο μεγάλες εσωτερικές ανισότητες. Η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα δεν είναι Τουρκία. Η Τουρκία είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Τώρα για τα δικαιώματα των α, ε, κουρδισών γυναικών. Ξέρω ότι εκεί ο ρυθμός των ε, γυναικών που είναι αγράμματες είναι πολύ ψηλός. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καν τη δική τους γλώσσα. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερες πληροφορίες. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των γυναικών των Κουρδισσών. Δεύτερο ερώτημα. Τα σημαντικά ποσά οικονομικής βοήθειας από ευρωπαϊκές χώρες. Και η χώρα μου συμβάλλει, συνεισφέρει οικονομικά. Αυτή η οικονομική βοήθεια που πηγαίνει κατά πόσο πηγαίνει για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίω των ΜΚΟ. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν ε, ευρωβουλευτές που, δια, που και βουλευτές Τούρκοι που διαμαρτύρονται ότι τα κονδύλια αυτά δεν πηγαίνουν στη βάση. Μια ακόμα ερώτηση. Αυτό που είπε προηγουμένω και η κυρία Γιανακουδάκη. Ένας από τους λόγους που οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις καθυστερούν, το είπε και ο κ. Σανίνο, είναι ότι η Τουρκία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της έναντι της Ένωσης. Για την Κύπρο, για παράδειγμα. Είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Δεν το έκαναν. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μια σειρά πραγμάτων που δεν έκαναν. Πώς μπορώ να πισθώ ως Ευρωβουλευτής ότι αυτά που υπόσχεται η Τουρκία για τα δικαιώματα της γυναίκας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα προστατευτούν πραγματικά και ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Ένωσης. Αν τόσο ζωτικές υποχρεώσεις όπως την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αναγνωρίστηκε εδώ και 7 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το ζητάμε από την Τουρκία κάθε χρόνο. Α, κάτι ακόμα. Υπάρχει μια, μια φράση που λέει ότι η συμμετοχή των γυναικών στους, σε κάποιους τομείς τραπεζικούς κλπ. είναι από, τις υψηλότερα, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η ερώτηση μου προς τον κύριο Σενίνο είναι σωστό γιατί εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Για μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Ehm, Ευχαριστούμε κύριε Παπαδοπούλου. Δεν βλέπω κανέναν άλλον που θέλει το λόγο. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη θεματική ενότητα θα δώσω το λόγο στους ομιλητές να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους στέθηκαν. Η κυρία Τζόσκουν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Evet, e, e, Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μετέθησαν και αν τυχόν παραλείψω κάποιες ε, ερωτήσεις, σας παρακαλώ πολύ να μου το πείτε. Η κυρία Μπόσκουρτ αναφέρθηκε στην βία κατά των γυναικών. Όντως το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Και ε, εμείς έχουμε δει ότι όντως τα επίπεδα βίας κατά των γυναικών είναι σημαντικά. Επομένως προσπαθούμε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ιδίως στα πλαίσια της νέας μας νομοθεσίας, για να προστατεύσουμε περισσότερο τις γυναίκες έχουμε αναλάβει τα μέτρα εκείνα τα οποία θα μας επιτρέψουν να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν προβεί σε εγκλήματα ή σε πράξεις βίας κατά των γυναικών. Όσον αφορά το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις νοοτροπίες μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και για αυτό το λόγο θέλουμε να καταρτήσουμε καλύτερα τους αστυνομικούς. Για ένα μήνα 23 αστυνομικοί παρακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης προκειμένου να καταφέρουν να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών. Όσον αφορά τώρα τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της υγείας, Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που μια γυναίκα απευθύνεται σε μια νοσοκομιακή υπηρεσία, σε ένα κέντρο περίθαλψης, η υπηρεσία αυτή άμεσα ασχολείται με την εν λόγω γυναίκα. Κάθε φορά επίσης που μια γυναίκα προσφεύγει σε ένα αστυνομικό τμήμα, προβλέπουμε ότι θα εισακούεται το αίτημά της αμέσως Επίσης σε κάθε περίπτωση θα καταγράφεται η μαρτυρία της ε, ε, γυναίκας αυτής και όταν διαπιστωθεί ότι το αδίκημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό, τότε η ε, γυναίκα αυτή θα μπορέσει να έχει πρόσβαση σε ένα κέντρο περίθαλψης, σε ένα κέντρο υποδοχής. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα τέτοια κέντρα στην Τουρκία. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα μπορεί καμία υπηρεσία να αρνηθεί μια τέτοια παρεχόμενη, μια τέτοια υπηρεσία στις γυναίκες. Υπάρχουν λοιπόν τα κέντρα αυτά περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών στις γυναίκες. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα κέντρα υποδοχής, ε, προβλέπεται και αυτό το σύστημα των καταφυγίων όπως ακούσατε. Έχει συναυθεί μια συμφωνία και έχει υπογράψει μάλλον η κυβέρνηση μια συμφωνία για τα επόμενα χρόνια και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα μπορούν να παίρνουν μαζί τους και τα παιδιά τους σε αυτά τα κέντρα υποδοχής. Δεν Αναφερόμαστε όμω μόνο στο ζήτημα των αστυνομικών αρχών ή των κέντρων υγειονομική περίθαλψης. Θέλουμε να καταρτήσουμε και τους δημοσίου υπαλλήλους. 1.800 δημόσιοι υπάλληλοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης. Ως προς αυτό συγκεκριμένα προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για την ισότητα των φύλων Πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών. Γνωρίζουμε ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ακόμα επιληθεί σε θεσμικό όμω τουλάχιστον επίπεδο χάρη στην βοήθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνη, του Υπουργείου Υγεία και άλλων συμβαλωμένων μερών. Υπάρχει πλέον ο κατάλληλο συντονισμό που μα επιτρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Αν δούμε επίση και τα στατιστικά δεδομένα, συνειδητοποιούμε ότι ε, οι νόμοι οι οποίοι εγκρίθηκαν και υλοποιούνται όντω εφαρμόζονται στην πράξη, μεταφράζονται σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και βλέπουμε ότι ε, κάθε χρόνο ο αριθμός των ε, προσφυγών μειώνεται Μάλλον, ο αριθμό των προσφυγών αυξάνεται, οι γυναίκες δεν φοβούνται πλέον να πάνε στο δικαστήριο και να καταγγείλουν την βία την οποία έχουν υποστεί. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, χάρη στο πρόγραμμα αυτό καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο. Η κυρία Μπόσκουρτ μας ρώτησε αν έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο το ταμείο αυτό το οποίο αποφάσισε να δημιουργήσει ο Πρωθυπουργό μας. Κοιτάξτε, στο δημοσιονομικό σύστημα της ε, Τουρκίας προβλέπεται όντως η δημιουργία ενός ταμείου για την καταπολέμηση της βίας. Δεν προβλέπεται μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό. Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνη και το Υπουργείο Παιδείας που ε, ασχολούνται με αυτό το πρόγραμμα και κάθε Υπουργείο προβλέπει μια συγκεκριμένη επιμέρους χρηματοδότηση. Οι πόροι αυτοί λοιπόν πηγαίνουν για αυτό το πρόγραμμα. Κάθε θεσμικό λοιπόν όργανο πρέπει να καλύψει τις υποχρεώσεις αυτές που απορρέουν από αυτό το γενικότερο πρόγραμμα καταπολέμησης της βίας. Επομένως, όντως έχει προβλεφθεί μια χρηματοδότηση, αλλά στον προπολογισμό του κάθε Υπουργείου ξεχωριστά. Η κυρία Μπόσκουρτ επίση αναφέρθηκε στις θετικές διακρίσεις ορισμένου τομεί, όντω αυτό συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο. Μπορώ να σας πω ότι οι θετικές διακρίσεις ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Στο AKP βλέπουμε ότι υπάρχουν 78 υποψήφιες, στο MHP 48 Αναφέρομαι στις υποψήφιες που έχουμε στους εκλογικούς καταλόγους, τα εκλογικά ψηφοδέλτια. Το BDP έχει περίπου 40% γυναίκες υποψηφίους και πιστεύουμε ότι τα αριθμητικά αυτά στοιχεία θα αυξηθούν. Τώρα όσον αφορά πάντα τις θετικές διακρίσεις, αυτή τη φορά στον τομέα της απασχόλησης και της παιδείας, προσπαθούμε να εισαχθούν όντω αυτέ οι θετικέ διακρίσει στου τομεί αυτού και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην εξέλιξη τη υλοποίηση αυτών των θετικών διακρίσεων. Η κυρία Κορέλσεν αναφέρθηκε στην προοπτική 2020 και πιο συγκεκριμένα στο ότι η διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως να, μάλλον, αν θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το καθεστώς των γυναικών. Η διαδικασία προσχώρηση τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη τη δεν αρκεί. Οι γυναίκες είναι πιο απαιτητικέ στην Τουρκία. Από το 2000 και μετά δούμε τη σχετική νομοθεσία. Βλέπουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή έχει συμβεί σε νομοθετικό επίπεδο έχει στόχο να προωθήσει τις ε, περισσότερες αλλαγέ, να επιφέρει κάποιε θετικέ εξελίξει. Υπήρχαν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν. Η ε, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την ε, Ισότητα των ε, Φύλων συνέβαλαν στο να, να πετύχουμε ένα καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία στην Τουρκία. Προφανώς η διαδικασία προσχώρησης της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στο να σημειωθεί πρόοδος. Στην Ευρώπη άλλωστε ζουν πάρα πολλοί Τούρκοι. Και αυτή η σχέση είναι πολύ σημαντική για την ε, Τουρκία. Είναι σημαντικό να δυναμωθεί η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και αναφερθήκαμε και στα κριτήρια της Κοπενχάγης Όσον αφορά λοιπόν τα κριτήρια αυτά και όσον αφορά τα κριτήρια για την απασχόληση και αυτά αποτελούν τμήμα των στόχων που έχει θέσει η Τουρκία και προφανώς θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα σχετικά αιτήματα. βλέπουμε μάλλον αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Τουρκάλες και τις γυναίκες κουρδικής καταγωγής. Σύμφωνα με τη Συμφωνία της Λοζάνης δεν υπάρχει μειονότητα αυτή και όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι είναι υπήκοοι πρώτης κατηγορίας υπήκοοι που βρίσκονται ε, ισότιμα στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά όσον αφορά την υγεία, την απασχόληση, όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Όσον αφορά λοιπόν την ισότητα των ευκαιριών, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Όλες αυτές οι υπηρεσίες ισχύουν για όλους τους πολίτες. Όσον αφορά τώρα την χρησιμοποίηση της κουρδικής γλώσσας, ναι, η κουρδική γλώσσα είναι γλώσσα η τουρκική γλώσσα είναι γλώσσα, η γλώσσα εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως και κάποιοι σταθμοί οι οποίοι εκπέμπουν στα κουρδικά. Η επίσημη όμως γλώσσα της χώρας είναι η τουρκική. Δεν είμαι κάποια πολιτική προσωπικότητα, δεν είμαι πολιτικός. Ως υπήκος όμως της Τουρκίας πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται σε καθεστώς κατοχής η Τουρκία μαζί με άλλες χώρες, τέλος πάντων η Τουρκία χρησιμοποίησε τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες. Όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τις γυναίκες στην Ήπεθρο. Προσπαθούμε να δώσουμε ίσε ευκαιρίε και ισότιμε υπηρεσίε σε όλε τι γυναίκε, είτε πρόκειται για τον γεωργικό τομέα, είτε πρόκειται για άλλου τομεί. Οι Υπηρεσίε αυτέ λοιπόν ισχύουν για όλε τι ε, γυναίκε και προβλέπονται κάποια προγράμματα κατάρτιση και τον γεωργικό τομέα. στον αφορά τώρα την ληξιαρχική καταχώρηση των γεννήσεων, τι ληξιαρχικέ πράξεις γεννήσεων, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα καταχώρησης των γεννήσεων. Θα πρέπει ε, να συνδέσουμε το ζήτημα αυτό με το ζήτημα της εκπαίδευσης. Έχει μηχανογραφηθεί πλέον το σύστημα, ε, καταχωρούνται όλες οι γεννήσεις και δεν υπάρχει καμία διάκριση προς αυτό όσον αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πόρους, ε, κρατικούς πόρους σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και διεθνείς πόροι οι οποίοι μεταφέρονται στις οργανώσεις αυτές και συμβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο στον προπολογισμό των οργανώσεων αυτών όσον αφορά την υλοποίηση των υφιστάμενων ακόμα και μελλοντικών προγραμμάτων και εμεί προφανώ συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τι μη κυβερνητικέ αυτέ οργανώσει. Θα ήθελα να ολοκληρώσω γιατί μου λέει η Πρόεδρο ότι πιέζει ο χρόνο. στην Τουρκία, όταν αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευση και κατάρτιση, κάθε φορά που μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στην απασχόληση, τόσο μειώνεται και το ποσοστό των εγκλημάτων τιμής. Θέλουμε λοιπόν να ελοποιήσουμε όλους αυτούς τους στόχους με χρονικό ορίστα το 2020. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και σεβόμαστε τη ζωή όλων των πολιτών στην Τουρκία. Ο κύριος Ανίνο θα απαντήσει σε ερωτήσεις τώρα. Θα είμαι συντομότατος γιατί δύο ερωτήσεις μου έκαναν. Η μία αφορά τον αριθμό των έργων για την κοινωνία των πολιτών. Δεν έχω εξαντλητικό κατάλογο των έργων που ολοκληρώθηκαν από το 2005 και μετά. Θα έλεγα ότι τα περισσότερα από τα μισά πάνε σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό, αυτό το στοιχείο πρέπει να το ελέγξουμε σε σχέση με τα άλλα προγράμματα και έργα που έχουν ανατεθεί. Εμείς θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Πρέπει να δω πρώτα όλο τον κατάλογο των έργων σε αυτόν τον τομέα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία των γυναικών σε συγκεκριμένους τομείς ευθύνης ε, εργατικού δυναμικού. Εδώ η κυρία Τζέρ που ε, είναι στην Τουσιάντ και στην ομάδα εργασίας για την ισότητα των φίλων μπορεί να απαντήσει καλύτερα στην ερώτηση. Ευχαριστώ εξ ονόματος όλης της Επιτροπής. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας που συμμετέσχουν σε αυτό το τμήμα, σε αυτό το μέρος της ε, ακρόασης και περνάμε στο δεύτερο μέρος κατά το οποίο θα μιλήσουμε με θέμα «Οι γυναίκες στην Τουρκία ως παράγοντες προόδου, μέτρα βελτίωσης και βέλτιστες πρακτικές». Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να καλωσορίσω δύο εμπειρογνώμονες που προσεκλήθησαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας σήμερα. Καλώς ορίζω πρώτα την κυρία Νουρ Τζέρ που είναι η πρόεδρος της Τουρκικής Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Ένωσης, της Τουσιάντ. Έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την ισότητα των φύλων στην Κωνσταντινούπολη. Ε, ένα θερμό καλώς ήλθατε λοιπόν και έχετε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτα, αγαπητά μέλη, αντιπρόσωποι, βουλευτές που ενδιαφέρεστε. Έχω έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 90 με 94 ε, συμμετείχα για τις διαπραγματεύσεις ε, ποσοστώσεων στην κλωστή Φαντουργία και ήμουν το 82 διερμηνέας όταν ε, ε, ίσχυσαν οι πρώτες ε, ποσοστώσεις στον τομέα των ενδυμάτων πήγα στην Επιτροπή Διαπραγματεύσεων και το 1996 όταν δημιουργήθηκε η Τελωνιακή Ένωση ήμουν επικεφαλής της, του κλάδου ενδυμάτων και χάρηκα τόσο πολύ είπα θα ξαναγυρίσω στην δουλειά μου τώρα που δημιουργήθηκε ένα νέο άνοιγμα και ελπίζω ότι τα επόμενα 15 χρόνια θα μπορούσαμε και εμείς να γίνουμε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, βέβαια δεν είναι το θέμα μας η ένταξη, αλλά επειδή ήμουν ιδρυτικό μέλος πολλών μη κοιό γυναικών, αυτή τη φορά πάλι ασχολούμαι με το θέμα της ισότητας των φύλων που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα στην Τουρκία σήμερα. Εγώ είμαι επιχειρηματίας κυρία Πρόεδρε. Δίσταζα πολύ αν θα έπρεπε να δείξω το μικρό φιλμ που φτιάξαμε στην Τουσιάντη αν θα έπρεπε να κάνω την ε, ομιλία μου. Έχοντας ακούσει τις ομιλίες θα ρισκάρω να δείξω το φιλμ που δημιουργήσαμε ως Επιτροπή Ισότητας των Φίλων... και υπόσχομαι ότι θα διαρκέσει 14 λεπτά, εγώ θα μιλήσω 6 λεπτά για να προλάβουμε με το χρόνο. Αν έχω την αδειά σας. Διαπραγματεύομαι δηλαδή να μου δώσετε πέντε λεπτά παραπάνω από το τέταρτο που δικαιούμαι για να κάνω αυτή την ομιλία και να δείξω και το φιλμ. Γιατί το φιλμ είναι πολύ σημαντικό και αφορά πολλά από αυτά που είπαμε σήμερα. Και πρώτη φορά στην ιστορία οι, οι λύσεις και οι συστάσεις δίνονται από άνδρες που επελέγησαν από διάφορους κύκλους της τουρκικής κοινωνίας και δείχνει αυτό τη μελλοντική μας πορεία. Γιατί αν δεν έχουμε την ανδρική υποστήριξη στα θέματά μας, δεν θα επιταχυνθεί η διαδικασία. Μου επιτρέπετε λοιπόν να δείξω πρώτα την ταινία, το φιλμάκι αυτό. Ε, είναι εύκολο να διαπραγματευτείτε σήμερα μαζί μου. Είμαι ενδοτική. Θα το δείξουμε λοιπόν. Μετά η, η, η παρέμβασή σας όμως θα είναι σύντομη, οπότε προχωρήστε για να δούμε το φιλμάκι.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 Ήχο δεν έχουμε, δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε. Ήχος, ήχος δεν ε, υπάρχει, αλλά μπορείτε ίσως να διαβάσετε τους υποτίτλους ή τα στοιχεία που δείχνει η ταινία. Can you read the subtitles? Ε, μπορείτε να διαβάσετε τους υπότιτλους. Σαν καλό.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 Ευχαριστούμε πολύ που μας το δείξατε αυτό το φιλμ. Και τώρα θα σας δώσω λίγα λεπτά, κυρία Γκέρ, αν θέλετε να σχολιάσετε το φιλμ. Ελπίζω να καταφέρατε να διαβάζετε τους υποτίτλους, γιατί ήχο δεν είχαμε, αλλά ό,τι μπορούσαμε να πούμε το είπαμε, οπότε εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Βέβαια, ο πρώτος φεμινιστής του 20ου αιώνα και μάλλον τα γκρουπ μας έδωσε δικαιώματα και θα πρέπει να ευχαριστήσω με την πρώτη γυναίκα που πραγματικά συνέβαλε στη χειραφέτηση των γυναικών στην Τουρκία, μια αξιοσέβαστη γυναίκα Επίσης κάναμε μια σημαντική έρευνα που απαντά στην ερώτηση της κυρίας Παπαδοπούλου. 295 μέλη της, ε, του ΣΙΑΝΤΑ απάντησαν στην έρευνα. Μέσα σε 10 χρόνια η συμμετοχή, μάλλον το ποσοστό των γυναικών στην Τουσιάντα ανέβηκε από το 25% σε 35%. Αρχικά η συμμετοχή στο Συμβούλιο ήταν 3% και μέσα σε λίγα χρόνια ανέβηκε στο 8% στην DCAD. Ψηλότερο από τον μέσο όρο της συμμετοχής γυναικών ε, στις άλλες επιχειρήσεις. Τώρα έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στην Ένωση. Όταν βελτιώνεται η εκπαίδευση, η συμμετοχή φτάνει και στο 70%. Δηλαδή φτάνει στο ποσοστό των ανδρών. Είχαμε κάποια θετικά στοιχεία από τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Και τώρα ε, γρήγορα θα σας δείξω τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η γονική άδεια θα πρέπει να ισχύει και για τους δύο γονείς στην άτυπη οικονομία που αναφέρθηκε θα πρέπει να ε, μειώσουμε το ποσοστό της άτυπης οικονομίας, επίσης ε, της ε, οικονομίας. Οι γυναίκες πρέπει να προβάλλονται και να επιμένουν ε, στον ιδιωτικό τομέα. Θα, αν υπάρχουν ερωτήσεις και δεν προλαβαίνω τώρα, μπορώ να τα πούμε μετά. Για τη συμμετοχή στο Κοινοβούλιο φαίνεται ότι η συμμετοχή θα είναι 20%. Η, η συμμετοχή των γυναικών θα αυξηθεί γιατί υπάρχει μεγάλη υποστήριξη μιας ε, πλατφόρμας γυναικών η οποία ε, έχει και εμάς μέλη και άλλες οργανώσεις που αυτή τη φορά σε μεγάλες πιέσεις ε, στους πολιτικούς και για την κοινή στρατηγική, την ευρωπαϊκή στρατηγική στην ε, Τουρκία. Θέλουμε να μειωθεί η διαφορά ανδρών γυναικών μέχρι το 2020 και να καταπολεμηθούν οι, όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών. Ευθυγραμμιζόμαστε με αυτή τη στρατηγική, αλλά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα στην Τουρκία. Παρόλο που έχουμε πολύ ε, καλά αποτελέσματα και λέμε στους πολιτικούς και στην κοινότητά μας ότι είμαστε η 16η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίω, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και θέλουμε να γίνουμε η δέκατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά είμαστε οι τελευταίοι σχεδόν σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ε, ανδρών γυναικών. Χρειαζόμαστε δραστικά μέτρα και μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας, Ιταλίας και Σουηδίας. Έτσι λοιπόν, ναι, οι γυναίκες ε, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους είναι ίσες, αλλά θέλουμε να εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι νόμοι και ως μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουμε βαρύ καθήκον και πολλή δουλειά να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω την ομιλία αυτή και να δείξω και το φιλμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Και τώρα προχωρούμε στην κυρία Χάνταν Κανκλαγιάν. Ε, καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε στην Επιτροπή. Η κυρία Καγκλαγιάν είναι η φυγήτρια στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Ε, είναι επίσης ειδική σε συνδικαλιστικά θέματα και στην οργάνωση εργαζομένων στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τομέα στην Άγκυρα. Ε, καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Όταν είναι κανείς ε, από τους τελευταίους ομιλητές σε μια μακρά ακρόαση, ε, αυτό αποτελεί ένα μικρό ρίσκο, ελπίζω να μην σας κουράσω θα μιλήσω για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των εμποδίων που έχουμε, την πολλαπλή, τις πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη συμμετοχή στην πολιτική. Αυτό είναι ένας από τους τομείς έρευνάς μου. Επίσης, ένα άλλο είναι ο εθνικισμός και συμμετέχω και εργάζομαι και σε ένα συνδικάτο που έχει πάνω από 100.000 μέλη στην Τουρκία και έχω ειδικευτεί σε θέματα γυναικών. Δραστηριοποιούμε επίσης το γυναικείο κίνημα και πολλές φορές εκπροσώπησα τις ε, Κούρδες γυναίκες. Η κυρία Τσοσκούν σας έδωσε κάποια παραδείγματα για την κατάσταση σήμερα. Η κυρία Τζοσκούν ανέφερε τα διάφορα μέτρα. Πράγματι, έγιναν μεγάλα βήματα σε νομοθετικό επίπεδο. Όντως υπήρξαν και πολλές πρωτοβουλίες με στόχο την ε, ισότητα των δύο φύλων και τη μείωση της βίας. Όπως όμως είπαν και άλλοι ομιλητές, δυστυχώς δεν έχουμε επιτελέσει στην πράξη μεγάλες πρόοδους. Για παράδειγμα, υπήρξαν νομοθετικές προσαρμογές στο θέμα βία κατά των γυναικών, αλλά ακόμα κάθε μέρα τρεις γυναίκες στην Τουρκία χάνουν τη ζωή τους διότι έπεσαν θύματα βίας ανδρικής. Ακόμα υπάρχουν πολλά καθημερινά προβλήματα. Οι γυναίκες δεν προστατεύονται επαρκώς. Μια γυναίκα ήθελε να εγκαταλείψει τον άνδρα της πρόσφατα και αντιμετώπισε πολλές απειλές και βία ζήτησε βοήθεια, αλλά δεν την βοήθησαν. Ε, και ο πρώην άνδρας της, ε, ενώ είχε, ήταν διαζευμένη, γι' αυτό δεν την βοήθησαν, και στο τέλος την σκότωσε ο πρώην σύζυγός της. Επίσης υπήρξε και η υπόθεση μιας 12χρονης η οποία ε, βιάστηκε από πολλούς άνδρες και η διαδικασία ε, στα δικαστήρια κράτησε μέχρι το 2010 από το 2003. Οι άνδρες γλίτωσαν με μια ελάχιστη ποινή. Παρόλη την κακοποίηση ε, που προκάλεσαν στο 12χρονο αυτό κορίτσι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τις ε, πρόοδους. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά ακόμη υπάρχουν πολλές αντιφάσεις, πολλά προβλήματα που δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποια είναι τα μεγάλα εμπόδια για μια αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των θεωρητικών βελτιώσεων. Καταρχήν, η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών προκύπτει από τις συμβάσεις και από τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάθε φορά ε, δεν ακολουθούμε μια συνολική προσέγγιση, ε, παρεμβαίνουμε εμβαλωματικά. Ας πούμε αυτή η θρησκευτική ε, συντηρητική ιδεολογία της οικογένειας που εξακολουθεί να υπάρχει και παίζει ρόλο. Από την άλλη προσπαθούμε να βάλουμε στην αγορά εργασίας τη γυναίκα. Ταυτόχρονα όμως ε, θέλουμε, την ενθαρρύνουμε να κάνει περισσότερα παιδιά, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Οι γυναίκες για να φροντίσουν τα παιδιά τους δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας. Η Μποσκούν το ανέφερε αυτό. Και πράγματι, στην Τουρκία δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Δεν υπάρχει υποδομή φύλαξης παιδιών. Οπότε... Δεν είναι ρεαλιστικό η γυναίκα να φροντίζει και τα παιδιά και την οικογένεια χωρίς τη βοήθεια του άντρα και να κάνει και σταδιοδρομία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εδώ και υπάρχουν και πολλά παραδείγματα ε, βίας. Τις περασμένες μέρες ένας ε, καθηγητής ε, θεολογίας έκανε δημόσιες δηλώσεις ότι οι γυναίκες πολλές φορές ευθύνονται για, την, για τις σεξουαλικές επιθέσεις, διότι προκαλούν τους άνδρες. Αυτό το πράγμα μπορεί να το πει ένα άτομο με μεμονωμένα. Είναι σημαντικό ποιο το λέει και είναι και σημαντικό τι συνέχεια δίνεται. Πώ αντιδρούμε. Τίποτα. Κανεί δεν είπε τίποτε. Δεν ε, λογοδότησε ο άνθρωπος αυτός ε, ούτε υπήρξαν ενστάσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα θεωρώ. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι και οι υπηρεσίες υγείας και, τις και οι υπηρεσίες ε, παιδείας ε, εμπορευματοποιούνται και θεωρούνται λιγότερο δημόσιο αγαθό. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι επίσης μια βασική προϋπόθεση για την ίση μεταχείριση. Αν δεν υπάρχει αυτό, πλήττονται οι γυναίκες πρώτες. Επίσης, ο μιλιταρισμός είναι σημαντικό ε, ανάχωμα για τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Όταν μιλάνε όπλα δεν ακούγεται τη φωνή των γυναικών. Τώρα, γιατί υποφέρουν πιο πολύ οι γυναίκες ε, Κούρδες. Είναι εκτεθειμένες σε πολυδιάστατες μορφές βίας Επί 40 χρόνια γίνονται ένοπλες συγκρούσεις, έχουν ξεριζωθεί χωριά, έχουν χάσει άνθρωποι πολύ τη ζωή τους και γυναίκες υφίστανται δεινά και επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Υπάρχουν σχετικές έρευνες με συμμετοχή ε, για τη συμμετοχή των ε, Κούρδων γυναικών στην ευημερία και ε, υποφέρουν και σε σχέση με τους άνδρες ε, ε, και πολιτιστικά. Η επίσημη γλώσσα τους είναι η τουρκική. Όταν πηγαίνουν οι άνδρες στο στρατό, ε, μαθαίνουν τουρκικά. Το γλωσσικό πρόβλημα για τις γυναίκες είναι μεγάλο όμως, γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Δηλαδή τα πολιτικά τους δικαιώματα δεν μπορούν να τα ασκήσουν επειδή υπάρχει ε, το εμπόδιο της γλώσσας για τις γυναίκες. Ε, οπότε χάνουν τα δικαιώματά τους ε, σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά αποτελούν διακρίσεις φύλου και βαθαίνουν τα προβλήματα. Επίσης, κάποια χωριά οπλίστηκαν για να προστατευθούν και έτσι αυξήθηκε ακόμη περισσότερο η βία κατά των γυναικών. Αυτό το σύστημα προστασίας των χωριών που εξοπλίζονται θέλω να το αναφέρω γιατί έτσι διαδίδονται πολύ τα όπλα και οι γυναίκες έτσι όχι μόνο υπόκεινται σε βία αλλά ε, φωνεύονται πολλές φορές γιατί ε, η βία γίνεται ένοπλη πια και είχαμε και περιπτώσεις αυτοκτονιών. που δείχνουν ότι οι γυναίκες ε, χρησιμοποίησαν τα όπλα εναντίον τους γιατί τα είχαν πρόχειρα. Ε, Επίση ε, πλήττονται πολύ από τους εκτοπισμούς στις περιοχές αυτές, ε, διώκονται οι γυναίκες. Πολλές φορές ε, αναγκάζονται να πάνε στις πόλεις, αφήνοντας τα υπάρχοντά τους εκεί και έτσι αυξάνουν το βαθμό εξάρτησής τους από την οικογένεια. πράγμα καταστροφικό. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες που πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. διότι οι δομές αυτές μεταφέρονται στις πόλεις ε, και ε, εξακολουθούν και διονίζονται εκεί. Και αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, η διάσταση της βίας ε, Α, οι εκτοπισμοί, ε, η αναγκαστική αστιφιλία, όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει η διάσταση του φύλου να περιλαμβάνεται σε όλους τους τομείς της πολιτικής και στους τομείς των εσωτερικών συγκρούσεων που υπάρχουν στην Τουρκία. Όλες αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να αναλυθούν και μέσα από το πρίσμα των γυναικών και αναζητώντας λύσεις θα πρέπει να αναπτύξουμε ιδιαίτερες πολιτικές υπέρ των γυναικών. Επίσης οι γυναίκες θα πρέπει να θεωρούνται ε, δραστήριοι, ενεργοί παράγοντες ε, στη διαδικα... στην προσπάθεια καταπολέμησης των διακρίσεων. Αυτό δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Αν δούμε το ρόλο των γυναικών σε όλους αυτούς τους τομείς, ε, βλέπουμε ε, πολλά προβλήματα και επίσης μπορούμε να εξηγήσουμε τα προβλήματα ε, των Κούρδων γυναικών και των γυναικών στην νοτιοανατολική Τουρκία δημιουργείται πολλές φορές ε, μία ε, διαφοροποίηση μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην Τουρκία. Δεν είναι όμως αυτές ε, οι περιοχές υπανάπτυκτες, είναι περιοχές που έχουν ταλαιπωρηθεί από συγκρούσεις, πόλεμες καταστάσεις και αυτή και μόνο η κατάσταση εξηγεί πολλά προβλήματα. Άλλωστε και στην Δύση βλέπουμε να μεταφέρεται η Ισλαμική κουλτούρα. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν πατριαρχικές δομές που πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι υπεραπλουστευτικό να ε, ε επικεντρωνόμεθα σε ορισμένους μονοτομείς, αγνοώντας πολλές φορές έτσι τα πραγματικά αίτια. Γιατί αν το κάνουμε αυτό περιθωριοποιούμε τους ανθρώπους και δεν βοηθάμε τις κούρτες γυναίκες που είναι θύματα βίας. Πολλές φορές δηλαδή θυματοποιούνται οι γυναίκες και ευθύς εξ αρχής ε, θεωρούνται ως θύματα. Ε, έχουμε τις προηγούμενες δεκαετίες ε, συλλέξει πολύ Πήρα από αυτούς τους τομείς και η πολιτική κινητοποίηση στις περιοχές των Κούρδων ε, ενίσχυσαν τις γυναίκες ιδιαίτερα ε, στον κοινωνικό και πολιτικό τους ρόλο. Μία έρευνά μου έχει ως αντικείμενο το κουρδικό και πώς επηρέασε το ρόλο των γυναικών και την ε, δραστηριοποίησή τους και διαπίστωσα ότι το πολιτικό κουρδικό κίνημα, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, αυτό το κίνημα λοιπόν, το πολιτικό, το κουρδικό, το επηρέασαν οι γυναίκες και το ε, ενίσχυσαν οι γυναίκες και μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποιήθηκαν οι γυναίκες και αυτό έδωσε εκπληκτικές επιπτώσεις ε, τώρα στην, ε, στο, ε, στο Κουρδικό Κόμμα έχουν εισαγάγει ποσοστώσεις και το 40% στα ψηφοδέλτια του 5P είναι γυναίκες και το 38% είναι εκλεγμένες ε, βουλευτίνες του Κουρδικού Κόμματος. Αυτό και τελειώνω τώρα δείχνει ότι μπορεί να υπάρξουν και αλλού παρόμοια παραδείγματα. Και πιστεύω ότι από την αρχή ε, το, αυτό που σημαίνει, αυτό που δείχνουν όλα αυτά είναι ότι πρέπει από την αρχή να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία οι γυναίκες. γυναίκες θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής να συμπεριλαμβάνονται. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και ζητώ από τις συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Η κυρία Μπόσκοτ πρώτη και καλύτερη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τις δύο εμπειρογνώμονες για τις παρεμβάσεις τους. Και έχω μια σειρά ερωτημάτων. Προς την κυρία Γκέρ. Χαίρο που βλέπω ότι οι επιχειρηματίες ε, έχουν σκεφτεί την συμμετοχή, την μείζωνα συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή της Τουρκίας ενώπιση του 2020. Συμφωνώ μαζί της ότι χωρί τις γυναίκε ανάπτυξη δεν υπάρχει. Άρα είναι προς και των γυναικών αλλά και των εργοδοτών και τη κοινωνία. Υπάρχουν πρωτοβουλίε συνεργασία με το κράτο. και αν ναι, πού βρίσκονται τα προβλήματα. Για την κυρία Τσαγκλάγια έρευνα. Είπατε ότι δεν υπάρχουν βελτιώσεις στον τομέα της βίας. Συμφωνώ μαζί σας, είχα επαφές πρόσφατα στην Τουρκία με πολλές γυναίκες που είναι και σε καταφύγια και μου είπαν σαφώς ότι οι χωρισμένες γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν ή να γίνουν δεκτές ακόμα και όταν ο πρώην σύζυγος της ε, ενοχλεί. Αυτό μου φαίνεται παράξενο διότι εκεί τότε χρειάζονται προστασία. Και με εντυπωσία του γεγονός ότι σε περίπτωση εμφανών ε, φαινομένων βίας μίλησε με μια γυναίκα η οποία είχε βασανιστεί, την είχε πιάσει στο δρόμο άντρας και την κλώτσαγε μετά τη... Ε, ε, τον χωρισμό. Τι έγινε. Έφτασε η αστυνομία, τον συνέλαβε τον ε, κράτησε για ένα 24 και μετά τον έστειλε σπίτι. Αν είχε κάνει ο άνθρωπος αυτός το ίδιο πράγμα στον γείτονά του, θα είχε γίνει μήνεση, θα είχε μπει φυλακή και θα είχε μια πολύ αυστηρότερη ποινή. Είναι λοιπόν σημαντικό να εφαρμόζονται οι νομοθετικές διατάξεις και να αποθαρρύνονται από τυχόν επανάληψη παρόμοιων εγκληματικών ε, στάσεων. Για την κυρία Τσαγκλαγιάν έχω ακόμα δύο ερωτήματα. Μιλήσατε για το 2020, τις προοπτικές του 2020. και για τα προβλήματα των Κουρδισών, των γυναικών από το Κουρδιστάν. Πώς μπορούμε αυτό το ειδικό ζήτημα να το ενσωματώσουμε στη στρατηγική ενόψη του 2020. Μια άλλη ερώτηση τώρα. Την περασμένη Δευτέρα απαγορεύθηκε η συμμετοχή ε, στους, στις εκλογές κάποιων γυναικών υποψηφίων από το Κουρδικό κόμμα πρόβλημα δημοκρατικό ευρύτερο. Είναι σημαντικό ο καθένα να μπορεί να κατέβει στι να εκλογέ. Τι άποψη έχετε από αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μπόσκουρτ. Η κυρία Κεστρελεύσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο φιλμάκι που είδαμε, είδε ότι οι γυναίκες στην Τουρκία είναι όχι μόνο 10% των βουλευτών, αλλά και σε άλλα επίπεδα τα νούμερα είναι χαμηλά. Και τούτο οφείλεται εν πολύ στην έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας. Οι γυναίκες της τουρκία έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν. Η κοινωνία ωστόσο βλέπει κάπως επιφυλακτικά τις εργαζόμενες γυναίκες οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας και μένουν τελικά σπίτι ή μένουν σπίτι για να ασχοληθούν με την οικογένειά τους. Όταν μπαίνουν στην αγορά εργασία συχνά υποχρεώνονται ε, να παραιτηθούν γρήγορα. Τα στατιστικά δείχνουν ότι στην αγορά εργασία η παρουσία της γυναίκας είναι αρκετά ασαφής. έλλειψη στην εκπαίδευση. Η έλλειψη στην εκπαίδευση έχει σημαντικές συνέπειες και πολιτικά και, οικονομικά. Παρά τα σημεία πρόοδου που αναφέρθηκαν υπάρχει υψηλότερο επίπεδο αναλφαβητισμού μεταξύ κοριτσιών και γυναικών και αυτό έχει αντίκτυπο και στην καθημερινότητα. Για μια ανγράμματη γυναίκα η δουλειά είναι πάντα πιο δύσκολα από ό,τι για τον άντρα. Επίσης, το θέμα της βίας και της ενδοοικογενειακής βίας, του είπε η κυρία Τσαγκλαγιάν. Το 39% των γυναικών που απάντησαν σε μία έρευνα σφίγγωμα μέτρησης δήλωσαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική βία. 4% όμως μόνο πήγε στην αστυνομία. Άρα, de facto, οι γυναίκες φοβούνται και γι' αυτό σιωπούν. Η θέση των γυναικών στην τουρκική κοινωνία κατά την άποψή μου συνεχίζει να είναι ασαφής. Η κυβέρνηση παρέχει εγγύηση ισότητας και στην αμοιβή και στην αγορά εργασία, στην πρόσβαση στην αγορά εργασία. Επί τη ουσία, ωστόσο και στις δημόσιε ακόμα θέσει, οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις. Η οικονομική ανεξαρτησία είναι σημαντική για τη χειραφέτηση της γυναίκας και η λειτουργία, αλλά η λειτουργία της κοινωνίας στηρίζεται ακόμα σε κάποιες αξίες παραδοσιακού χαρακτήρα και όχι στην νομοθεσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο νόμος είναι καλός, η πράξη είναι διαφορετική. Άρα ε, μάλλον οι γυναίκε χρειάζεται να αγωνιστούν συνεχώ για να δηλώσουν ε, την παρουσία του στην κοινωνία και η σύγκρουση μεταξύ νεοτερισμού και παραδοσιακών αξιών οδηγεί και, στην, και στον αγώνα για μια αξιοπρεπή ζωή. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό μόνο νομικά. Χρειάζεται και κοινωνική και νομική παρέμβαση. Όλο και καλύ... βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση ότι όλο και περισσότερε οργανώσει γυναικών εμφανίζονται που ζητούν όχι μόνο την εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και την εφαρμογή των διεθνών στάντα για τα δικαιώματα των γυναικών. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι καλύτερες είναι το τομέα της εκπαίδευσης. Αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξουν δράσεις εκτεταμένη, σε πιο εκτεταμένη κλίμακα ευαισθητοποίηση των γυναικών για τη, τα δικαιώματά τους. Και αυτό δεν αρκεί να περάσει μέσω νομικών πράξεων, αλλά και μέσω της επίγνωσης ότι η έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών οδηγεί σε σημαντικές σοβαρές συνέπειες. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνουν αποτελεσματικές δράσεις nie da się polecieć w przyszłość na jednym skrzydle. στο φιλμάκι ότι το μέλλον δεν μπορείς να το βελτιώσεις με ένα βήμα. Αλλά θέλουμε πολλά. Ρωτώ, πότε λοιπόν θα έχουν δύο φτερά οι Τουρκάλες για να μπορέσουν να πετάξουν προς ένα καλύτερο και πιο ε, ονειρεμένο μέλλον. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Παπαδοπούλου παρακαλώ. Με εντυπωσίασαν αυτά που άκουσα από την κυρία Τσαγκλαγιάν. Ξέρω την κατάσταση των ε, κουρδισών γυναικών και ήσασταν πολύ έντιμοι, παρουσιάσετε τα πράγματα όπως ήταν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Βλέπω από το προφίλ σας ότι είστε συγγραφέας, ακτιβίστρια, δουλεύετε για την ειρήνη, για το φεμινισμό, κατά των διακρίσεων ε, φύλου. Ρωτώ λοιπόν, σε τι βαθμό μετέχετε στις συζητήσεις, στο κοινωνικό διάλογο, με εκπροσώπηση των γυναικών από το Κουρδιστάν. Όταν είχα πάει στην Τουρκία, ρώτησα, συμμετείχαν οργανώσεις γυναικών στον κοινωνικό διάλογο για τις ε, αλλαγές και στη συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε, ακούστηκε ένα παράπονο ότι δεν υπήρχε ενεργή παρουσία εκπροσώπων από το Κούρδισταν αλλά και από και κάποιον ΜΚΟ. Εσείς μετέχετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας σας. Δεύτερον, το μαζικό δημοκρατικό έλλειμμα που είπατε ότι υπάρχει ακόμα. Πιστεύετε, είστε αισιόδοξοι, θα υπάρξει αλλαγή. Τα εμπόδια που αναφέρατε θα αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένη στρατηγική. Βλέπετε βούληση της τουρκικής κυβέρνησης να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά και να δώσει πραγματική εξουσία στις γυναίκες. Και ένα σχόλιο στην κυρία Κοσκιούν. Είπε ότι δεν είναι πολιτικό, αλλά είπε ότι δεν υπάρχει εισβολή στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι σωστό. Θέλω να ρωτήσω μια Κούρδισσα που υποφέρει λόγω της καταστολής των δικαιωμάτων, τη καταπίεσης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Τουρκία. Κατά πόσο υπάρχει κατοχή ή όχι στην Κύπρο. Διότι ξέρω πως υπάρχουν τουρκάλες γυναίκες που υποφέρουν στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου Πρόσφατα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τώρα ακόμα γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις όπου μετέχουν γυναίκες του κάλες που διαμαρτύρονται για την κατοχή της Τύρκου στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Και εγώ δεν είμαι πολιτικό ζώο, είμαι μια γυναίκα που αγωνίζομαι για τα δικαιώματά μου. Ευχαριστώ κύριε Παπαδοπούλου. Για ένα λεπτό η κυρία Τέκιν. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις για την κυρία Γκέρ. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τους, την, τους επιχειρημα, την επιχειρηματική κοινότητα της Τουρκίας της Βρυξέλλες. Επιχειρηματικά. Δηλαδή από την οπτική αγωνία της επιχειρημα, των επιχειρηματιών. Πώς μπορεί να βελτιώσουμε τα επιχειρηματικά εργαλεία των γυναικών στην Τουρκία. Δι, δεύτερον, τα, οι μακροπιστώσεις, όχι οι μικροπιστώσεις. Οι μικροπιστώσεις υποστηρίζουν τις φτωχές γυναίκες για την καλύτερη ανάπτυξη συστημάτων μακροπιστωτικών ε, δανείων στην Τουρκία. Τι έχετε να πείτε. το 10% που είναι όριο για να περάσει κανείς στη Βουλή, εσείς μιλήσετε για, τα, για τις ποσοστώσεις, το 10% που έχουν οι Τούρκοι για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου να θέλουν το λόγο. Θα δώσω το λόγο στο πάνελ των προσκεκλημένων μας για να απαντήσουν. Πρώτα πρώτα κυρία Γκέρ. Um, Ευχαριστώ. Για την κυρία Μπόσκουτ Πώς συνεργαζόμαστε με τις κυβερνητικές αρχές για τη βελτίωση της κατάστασης. Το φιλμάκι έγινε γιατί θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για την κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία. Όταν είδαμε την πραγματική ζωή καταλάβαμε ότι για να μπορεί η γυναίκα να μπει στον κόσμο των επιχειρήσεων θα έπρεπε να βελτιώσουμε το σύστημα νηπιαγωγείων, βρεφονηπιακών σταθμών και παιδικής μέρημνας γενικότερα. Γιατί ο μόνος, μόνο, γιατί μια γυναίκα θα αρχίσει να δουλεύει μόνο αν έχει καλή ε, προστασία, καλή μέρημνα των παιδιών. Και ετοιμάζουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που θα υποβάλουμε στην ε, μετεκλογική κυβέρνηση με τίτλο «Ένας παιδικός σταθμός» Πώς το λέμε το κρέσ στα αγγλικά, λέει ο Μιλήτρια. Ένα λοιπόν υπηαγωγείο, παιδικός σταθμός, ένας παιδικός σταθμός σε κάθε δρόμο massive uh, project uh, to uh, Προωθούμε αυτή την ε, ιδέα για να μπορέσει εύκολα κάθε γυναίκα να έχει δυνατότητα να αφήσει το παιδί της και να πάει στη δουλειά της. Πρωτοβουλίες είναι αυτές. Επίσης δουλεύουμε με μια άλλη ιδέα. Παραμάνες ημέρας κάποιες γυναίκες να φροντίζουν αφού περάσουν από κάποια εκπαίδευση ε, τα παιδιά εργαζόμενων γυναικών. Τρίτο σχέδιο που απαιτεί νομοθεσία. Όχι νομοθεσία, προσε, διαφορετική προσέγγιση. Ξέρετε, στην Τουρκία πάει ο κόσμο καινούριε οικιστικέ περιοχέ με 5 10000 ανθρώπου. ανθρώπους. Οπότε ε, θέλουμε νομοθετικά κάθε καινούριο οικισμό να περιλαμβάνει παιδικό σταθμό ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού. Αυτό θα κάνουμε, θα προτείνουμε στις κυβερνήσεις για να διευκολύνουν ε, τη ζωή των εργαζόμενων γυναικών. Να πω όμως και κάτι για την κοινωνική κατανόηση. Το 62% των γυναικών αποκαλούν αυτές νοικοκυρές. σε αντιδιαστολή με τις γυναίκες που κάνουν σταδιοδρομία, σαν να μην είναι σταδιοδρομία ή το να είσαι νοικοκυρά. Όταν τους ρωτάμε θέλετε να δουλέψετε, οι δουλειές υπάρχουν, μισθοί υπάρχουν, συνεχίζουν πολλές γυναίκες να λένε ότι δεν θέλουν. Θέλουμε λοιπόν να προσφέρουμε τα κίνητρα, ούτως ώστε οι γυναίκες να το θέλουν να πάνε να δουλέψουν και να έχουν οικονομική ανεξαρτησία. Αλλά από την άλλη μεριά πολλές απόφοιτες πανεπιστημίου συνεχίζουν, αποκτούν, πηγαίνουν στην αγορά εργασία, δουλεύουν 70% και δουλεύουν και συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμα και αν κάνουν μέχρι δύο παιδιά. Τώρα, για το ερώτημά σας μικρο-μάκρο πιστώσεις. Η Κέργκινταρ, η οργάνωση, η οργάνωση που εκπροσωπείται, έχει ένα πρόγραμμα τριετές ε, πηγαίνουμε σε, με μια, συνεργαζόμαστε με μια ιδιωτική τράπεζα και πηγαίνουμε σε κάθε πόλη δημιουργώντα κίνητρα για επιχειρηματικότητα, προσφέροντα εκπαίδευση στις γυναίκες να γίνουν επιχειρηματίες. Και πάλι, ωστόσο, πολύ μικρό ποσοστό γυναικών είναι επιχειρηματίες στην Τουρκία. Τι, δεν χρειάζεται να σα το πω, με 20% αναλφαβητισμό μεταξύ των γυναικών, και με ένα μικρό ποσοστό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μεταξύ των γυναικών, είναι δύσκολο. Για να γίνεις επιχειρηματίας πρέπει πρώτα να δουλέψεις, να αποκτήσεις τεχνογνωσία, παιδεία και μετά να γίνεις επιχειρηματίας. Γι' αυτό η γυναίκα δεν έχει... Δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία της γυναίκας στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Πριν λοιπόν ε, τα δάνεια πρέπει να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ισότητας στη γυναίκα. Και ξέρετε, τα μέσα στην Τουρκία δεν, δεν επιτρέπουν στη γυναίκα να εμφανίζεται πραγματικά ίση. Σαν ΜΚΟ εμείς ε, προσπαθούμε να δουλέψουμε για να επιταχύνουμε την ε, ισότητα. Και ξέρετε στην πολιτική είχαμε μια πολύ καλή ε, συμμετοχή, μια σημαντική παρουσία γυναικών στη Βουλή, 120 γυναίκες. Πρώτη φορά στην ιστορία μας. Και αυτό επιτάχυνε και την νομοθετική παραγωγή και απαιτέλεσε παράδειγμα για το μέλλον. Κοιτάξτε, ένα νερό όταν βάζουμε το νερό να βράσει θέλει πολύ ώρα για να βράσει αλλά αρχίζει κάποια στιγμή να βράσει. Εμεί στην Τουρκία πήγαμε γρήγορα. Παρότι τα νούμερα σήμερα δεν είναι επιβοηθητικά, αλλά για μένα τα νούμερα αυτά δείχνουν το παρελθόν. Εγώ πιστεύω ότι σύντομα θα προχωρήσει η ε, ενδυνάμωση των γυναικών πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ κι εγώ. Κύριε Τσάγκλαγιαν. Ευχαριστώ. για το όριο συμμετοχής των κομμάτων στη Βουλή, το 10%. Αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνη, είναι ένα σαφές εμπόδιο στη δημοκρατία. Αυτά για το θέμα αυτό. για την απαγόρευση των μελών του BDP, γυναικών ή ανδρών. Να σας πω ότι στο BDP οι γυναίκες έφτασαν σε ένα επίπεδο εκπροσώπησης που, που για την Τουρκία είναι μοντέλο. Θετικό μοντέλο. Και αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Διότι οι γυναίκες που είναι στο κόμμα αυτό είναι μεσαίων τάξεων, μάλλον εκπαιδευμένες, εν γέννη. Ωστόσο, στο 5P οι γυναίκες προέρχονται από τελείως, διαφορετικό, ε, από διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Όταν βάζουμε εμπόδια λοιπόν στην παρουσία αυτών των γυναικών στην πολιτική, δημιουργούμε κοινωνιακά προβλήματα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες κουρδικής προέλευσης, αλλά τις γυναίκες γενικότερα. Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή οι γυναίκες από το Κουρδιστάν, οι φεμινιστικές οργανώσεις, έχουν ξεκινήσει έναν επικοδομητικό διάλογο που λειτουργεί καλά, πολύ καλά. Με σαφή αμφίδρομο χαρακτήρα. Η συνεργασία των γυναικών δεν γίνεται μόνο γίνεται ούτω ώστε η κοινωνική ειρήνη να υλοποιηθεί στην πράξη και να υπάρξει μάχη πραγματική αντιμετώπιση του αποκλεισμού οργανώσεις των γυναικών συζητούν μια σειρά θεμάτων. Η πρωτοβουλία των γυναικών για την ειρήνη, για παράδειγμα, ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από γυναίκες και στην οποία μετέχουν γυναίκες από διάφορα κόμματα της Τουρκίας. Είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να υποστηρίξουμε. Τώρα, για τον κοινωνικό διάλογο κάποια βουλευτής με ρώτησε για τη συμμετοχή μου στον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο πιστεύω ότι η γενική κατεύθυνση για την κατάσταση των γυναικών ε, με, με, μου κάνει να συμμετάσχω σε μια τέτοια συνάντηση. Τώρα, σε εθνικό συνδικαλιστικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, να σα πω ότι δεν έχω συμμετάσχει ακόμα σε καμία, σε καμία, διεθνή, σε καμία διεθνή δομή. Μου τέθηκε επίσης το ερώτημα κατά πόσον εν ώψη όλων αυτών των ανητικών στοιχείων που περιγράψα, αν έχω ελπίδες. Ναι, έχουμε κερδίσει μάχε. Έχουμε αποκτήσει κάποια κεκτημένα, όπω αυτή του 2005 ε, υιοθετήθηκε το πέντε ένας νέος αστικός κώδικας. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν πολύ για να αλλάξει ο αστικός κώδικας. Και η ενταξιακή διαδικασία είναι σημαντική, αλλά το γεγονός ότι βγαίνουν οι γυναίκες στο δρόμο και αγωνίζονται για, κάποια, για κάποιους στόχους Πιστεύω ότι αυτό θα προχωρήσει τα πράγματα και θα προχωρήσει και την εμπειρία τους. Νομίζω ότι απάντησα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπήρχε και μία ερώτηση προς την κυρία Τσόσκουν. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ένα ζήτημα. Η κυρία Μπόσκουρτ είπε το ακόλουθο. Αναφέρθηκε σε αυτά τα κέντρα υποδοχής, αναφέρθηκε στις γυναίκες εκείνες οι οποίες δεν χαίρουν προστασίας μετά από διαζύγιο. Έχει εγκριθεί όμως μία νομοθεσία, η υπαριθμών 1320, που έχει ως στόχο την προστασία της οικογένειας. Αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι πολύ συχνά ότι ο σύζυγος είναι αυτός που είναι βίαιος και προβλέπει η νομοθεσία αυτή την απομάκρυση του βίαιου συζύγου από τη σύζυγο. Και κατά αυτόν τον τρόπο η σύζυγος έχει και τη δυνατότητα πιο ήρεμα να απευθυνθεί στην αστυνομία ή σε υγειονομικές υπηρεσίες. Ο ποινικό πάντω κώδικα δεν προβλέπει μια διάκριση ανάμεσα στι έγγαμε ή διαζευγμένε γυναίκε. Όσον αφορά λοιπόν την επίθεση, τη βία ή την παρενόχληση, ο υπέτειος είναι αυτός ο οποίος καταδικάζεται, είναι το άτομο στο οποίο επιβάλλονται οι κυρώσεις. Η νομοθεσία λοιπόν για την προστασία της οικογένειας θα τροποποιηθεί οποιοδήποτε και να το καθεστώ των γυναικών, έγγαμοι, μη παντρεμένοι, διαζευγμένοι, απλώς αραβωνιασμένοι, οποιοδήποτε και να το καθεστώ στις γυναίκες θα μπορεί να χαίρει από την προστασία την οποία της προσφέρει πλέον ο νόμος απέναντι στον σύζυγο ο οποίος υπήρξε βίαιος. Όσον αφορά τα παιδιά, ιδίως για αυτά που βρίσκονται μεταξύ τριών και 5 ετών, Βλέπουμε ότι είναι όλο και περισσότερα αυτά τα οποία είναι ενταγμένα στο σχολικό σύστημα και καταβάλλονται πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο κατάρτισης, το επίπεδο εκπαίδευσης και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες θα συμμετέχουν στην αγορά, στην αγορά εργασίας. Μου τέθηκε ένα ερώτημα όσον αφορά τις μελλοντικέ προοπτικές. Τα μαθήματα τα οποία διοργανώνονται για την βελτίωση του επίπεδου κατάρτισης ε, των γυναικών, όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την βελτίωση της κατάστασης της γυναίκας, προβλέπουν μία κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου με συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος και πάλι εδώ είναι οι γυναίκες να έχουν όλο και καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θέλουμε λοιπόν να θέσουμε νέους στόχους, έχουμε πλέον ένα νέο όραμα και θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας αυτούς. Το όραμα θα γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μπόσκουρτ, για να συνοψίσει τη σημερινή μας απογευματινή συζήτηση. Έχετε το λόγο, κυρία Μπόσκουρτ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση, αυτό το οποίο μου ζητάτε, να καταφέρω να συνοψίσω την απογευματινή μας συζήτηση. Οι περισσότεροι πάντως υπογράμμισαν, τόνισαν ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην ομοθεσία από τη μια και την, τα όσα συμβαίνουν στην πράξη από την άλλη. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε στην υλοποίηση, την εκτέλεση των νομοθεσιών που έχουν εγκριθεί στην Τουρκία. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα γυναίκες οι οποίες είναι θύματα βίας και στο μέλλον το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακρινό μέλλον τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Η Τουρκία δεν μπορεί να προοδεύσει χωρίς τις γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες. Πρέπει να αλλάξει η αγορά εργασίας, πρέπει να προοδευσει όλε οι απαραίτε πρεπει λοιπον να καταβληθουν ολε οι απαραιτητες προσπαθειες πρεπει να αλλαξει η αγορα εργασια πρεπει να αλλαξει το σύστημα κοινωνική ασφάλισης, το σύστημα φροντίδα για τα παιδιά σε όλου αυτού του τομεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι ένα 20% μόνο των γυναικών αυτό που έχει πρόσβαση στην αγορά εργασία. Προκειμένου όμω να δουλέψουν περισσότερε γυναίκε, πρέπει να αυξηθεί η πρόσβασή του, πρέπει να δημιουργηθούν θέσει εργασία και παράλληλα πρέπει να δημιουργηθούν όλε οι συμπληρωματικέ υπηρεσίε που θα τι βοηθήσουν να αφήσουν το σπίτι. Δηλαδή η παιδική σταθμή, οι υπηρεσίε φροντίδα των παιδιών, Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση γιατί διαφορετικά οι γυναίκες δεν θα καταφέρουν να βγουν από το σπίτι, δεν θα καταφέρουν να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα θετικής διακριτικής μεταχείρισης κάθε φορά που εντοπίζουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Το Σύνταγμα πλέον επιτρέπει τις αλλαγές αυτές, επομένως δεν υφίσταται πλέον η δικαιολογία αυτή. έγιναν οι απαραίτητε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και αυτό μάλιστα με πολύ μεγάλη συνένεση του τουρκικού πληθυσμού. Ξέρετε ότι είχαμε ένα δημοψήφισμα, ότι έγινε ένα δημοψήφισμα τον Σεπτέμβριο. Εναπομένει λοιπόν, εναπόκειται πλέον στην κυβέρνηση να προβλέψει πλέον τι απαραίτητε νομοθεσίε, του απαραίτητου νόμου και κυρίω την εφαρμογή των νόμων αυτών προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση. Νομίζω ότι η σημερινή μα ακρόαση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε τα εφιστάμενα προβλήματα. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας επίσης στα υφιστάμενα προβλήματα τα οποία έχω εντοπίσει στην έκθεσή μου, προκειμένου να έχουμε πραγματικά μια προοπτική του 2020 για τις γυναίκες στην Τουρκία. Πρέπει καταρχάς να εστιαστούμε στα σημερινά προβλήματα. Με, τις συναδέλφους μου, λοιπόν, με τους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εστιαστούμε στα προβλήματα αυτά προσπαθώντας όμως να δημιουργήσουμε και ένα υψηλότερο επίπεδο ελπίδας και αισιοδοξία για την αυτονομία των γυναικών στην Τουρκία. Αυτά μπορούμε να κάνουμε για τις γυναίκες στην Τουρκία, αυτές τις συγκεκριμένε προτάσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα, με την συνεργασία λοιπόν των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τις τουρκικές αρχές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Τουρκία θα καταφέρουμε πιστεύω να πετύχουμε το στόχο αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους, στις προσκεκλημένες ε, εμπειρογνώμονες που ήρθαν και παρουσίασαν την εμπειρία τους. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους και όλους όσους συμμετέσχουν και τη γραμματεία προφανώς που μας επέτρεψε να οργανώσουμε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε και ε, να σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ.